and Mr. David. You can invite me for a beer afterwards, but now we will vote. He doesn't listen to you. No. We will start with... Ας αρχίσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες με την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Βάιντερ. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Βάιντερ. Ναι, αλλά ακόμη μπαίνει ο κόσμος. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, μου επιτρέπετε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε με τους ενδιαφερόμενους. Πολύ πρωτότυπο αυτό το θέμα, πολύ καινοτόμο και Χάρηκα ιδιαίτερα που ανέλαβα αυτή την έκθεση. Είχαμε 124 τροπολογίες, απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντος που προκάλεσε η έκθεση στους συναδέρφους. Χάρη σε αυτές βελτιώθηκε η έκθεση και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω εκ βάθος καρδίας τον κύριο Μάρτιν, την κυρία Σάκε, τον Ρούι Ταβάρες, τη Μαρή Κριστίν Εντζιάρ και τον Τσάρ Στάνοκ για την ανεκτήμητη συνεισφορά τους και την ορατή βελτίωση της έκθεσης στην οποία συνέβαλαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ανάπτυξης, γιατί πολλά από τα σημεία της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, περιλήφθηκαν ε, στις τροπολογίες των συναδέλφων και σωματώθηκαν στην έκθεση. Ευχαριστήσω λοιπόν και ε, την κυρία Μπόμπιτς και την κυρία Πάτης για την μεγάλη τους βοήθεια. Στόχος έκθεση ήταν να βρούμε απτές λύσεις τα πιο κατεπήγοντα προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι πεπισμένη ότι τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ.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 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος. Την 101. <laughs> Die Πέρα ψηφοφορία. geschlossen. ψήφοι υπέρ και δεν έχω την ε, κάρτα μου μαζί και ψηφίζω υπέρ όπως και οι σοσιαλιστές. Δεν έχουμε σοσιαλιστές, μόνο Ευρωπαίους έχουμε. 30 ψήφοι υπέρ λοιπόν και 27 κατά. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Εκατόν τέσσερα λοιπόν λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά Να το ελέγξουμε, αν και μου φαίνεται ότι έγκρινεται με την ίδια πλειοψηφία. Την 108 παρακαλώ, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. τη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 42 κατά. Απορρίπτεται. Εκατόν εννέα υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά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 για την 115. Πέρα ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 και 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, συγγνώμη 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος ζητείτε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 30 υπέρ, 29 κατά. Μα το ήξερα, σας το είπα. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε παρακαλώ. Αν συμμετέχετε όλοι, είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Αλλιώ όταν είναι οριακό το αποτέλεσμα είναι δύσκολο. For against. Which report? Uh, let's see the American Express. 58, there's one too many. Oh, no, it's okay now. Η Abstimmung ist geschlossen. Βλέπετε πόσο σημαντική είναι η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 44 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Εντάξει. Abstimmung ist geschlossen. Πέρα 32 υπέρ, 34 κατά απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 41-42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Die Abstimmung ist geschlossen. ψήφοι υπέρ, 30 κατά εγκρίνεται. Η 43 τώρα. Καταπληκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά αποχές Ξανά για την 8 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται 31 ψήφι υπέρ 35 κατά. ΔΕΒΕ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ΔΕΒΕ 2 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται ΔΕΒΕ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Εδώ στη μέση δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας. Πέρα ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 46 κατά απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Να το ελέγξουμε παρακαλώ, δεν είμαι σίγουρος. Για την ΤΕΒΕ 12. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα φορέας 34 τέσσερις υπέρ, τριάντα κατά εγκρίνεται. Μην ΤΕΒΕ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΤΕΒΕ 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, έλεγχος. Πέρα ψηφορίας. 25 ψηφοί υπέρ, 41 κατά, απορρίπτεται. 20 μέχρι 25 να τις ψηφίσουμε μαζί. Μάλιστα, συμφωνείτε. Υπέρ για την 20 έως 25. Όχι. Χωριστά. Η 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. 47 ψήφι. υπέρ, 3 κατά, 17 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση και συγχαίρω την κυρία Διακόμνουν. Και τώρα περνάμε στην έκθεση για την Κροατία. Ο Ρίβορ Ρούτσεκ είναι ο μας. Έχετε να πείτε κάτι. αν όχι να αποφανθούμε κατευθείαν. Τέσσερα. Τροπολογία τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επτά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εννέα. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δέκα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Μάλιστα, έλεγχος. Πέραση της ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12-13 υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Του συγητή. Α, συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 27 υπέρ. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία προφορική τροπολογία να κάνω μετά τη συμβαστική 2 να τη διαβάσω. Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνεργασία με τις αρχές της Κροατίας σε φάσεις ε, μετά την ένταξη και υπογραμμίζει ότι μια τέτοια, ένας τέτοιος μηχανισμός εποπτείας είναι ε, βασικός για να διασφαλίσει την ε, βιωσιμότητα των εργαλείων κατά τη οργανωμένου εγκλήματος και τονίζει ότι αυτό θα αποβεί σε όφελος των κρατικών αρχών και των κρατών πολιτών προκειμένου να συνεχιστούν και οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το κείμενο που προτείνω. Να σας πω, γιατί κατατίθεται ως προφορική τροπολογία, συμπεριλήφθησε ε, στις γραπτές ε, τροπολογίες που δεν καλύφθηκε από την συμβαστική 2. Θεωρήθηκε ότι καλύπτεται, αλλά δεν θεωρώ ότι καλύπτεται. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να ψηφιστεί. Ο εισηγητής. Πρόεδρε, Είμαι κατά του μηχανισμού εποπτείας μετά τις 1 Ιουλίου για την Κροατία. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο δική μου άποψη, αλλά είναι και η άποψη των σκιωδών. Ωστόσο, αν η κυρία Μακοβέη επιθυμεί να την ψηφίσουμε, ας την ψηφίσουμε. Ο κυρία Νέιτς. Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Δέχομαι την ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλίας για ε, όλους τους συναδέλφους, αλλά η συζήτηση έληξε χτες και τώρα η κυρία Μακοβέη θέλει να επανέλθει στο θέμα υπό μορφή ε, προφορικής τροπολογίας. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Γι' αυτό θεωρώ ότι παρόλο, παρόλα όσα είπε ο κύριος Ρότσεκ θα πρέπει να απορρίψουμε την τροπολογία. Δεν μπορεί κανείς να συνεχίζει επί μακρόν στο δινεκές. Είπατε ότι είσαστε κατά της ψηφοφορία λοιπόν κυρία Νέιτς. Είπα ότι δεν θα προτιμούσα να ψηφίσουμε τώρα. Αν θέλουν οι συνάδελφοι οπωσδήποτε να ψηφίσουν, εγώ απλά αναφέρω ότι δεν είναι τρόπος ε, να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν πρέπει να πάρει ποτέ τέρμα η συζήτηση. Απάντηση εκτός μικροφώνου. Κυρία Μακοβέη, λέει ο Πρόεδρος. Αν ένα μέλος αντιταχθεί στην ψηφοφορία, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Αυτοί είναι οι κανόνες. Δεν κατατίθεται όμως επίσημη ένσταση, άρα ας ψηφίσουμε. Ο κύριο Αλαφράγκα. Πρόεδρε, θα πρέπει να διασαφηνίσουμε αυτό το θέμα το διαδικαστικό και δεν αναφέρομαι σε μια προφορική γιατί δεν θα πρέπει να είμαστε ανέλικτοι. Θα πρέπει η πλειοψηφία της Επιτροπής να αποφανθεί. Θα πρέπει όμως να μας διέπει ένα δόγμα, μία αρχή, όπως είναι η περίπτωση αυτή. Προσωπικά πιστεύω ότι ότι ο συμβασμός είναι ασύμβατος με την πρόταση συμβασμού. Εάν το επιθυμείτε όμως, μπορούμε να αποφανθούμε και νομίζω ότι θα αποφανθούμε κατά. Θα διαγραφεί μια πλειοψηφία κατά. Κύριε Σαλαφράγκα, ακριβώς αυτό προτείνα. Δεν κατατέθηκε επισήμως ένσταση. σε ενδεχόμενη ψηφοφορία, άρα θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ ποιο είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας της κυρίας Μακοβάη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 ε, υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά άποχες. Ε, θεωρώ ότι εγκρίνεται, αλλά να κάνουμε και ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Die Abstimmung Πέρας ψηφορίας. 37 υπέρ, 27 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην 56. Ε, Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Στο δεύτερο τμήμα γιατί το πρώτο καταπίπτη, εφόσον εγκρίθηκε η συμβαστική 5. «56, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 55, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 60, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Κατά πάσα πιθανότητα εγκρίνεται. Ελέγχουμε. 61. Για την 61. Πέρας ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ, 32 κατά, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Οι 2 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Και τώρα παγκρινάμε στη συνολική ψηφοφορία υπέρ της έκθεσης ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας 60 ψήφι υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Συγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στην κύριο Ρούτσεκ. Να δούμε αν θα σημειώσει παρόμοια επιτυχία και ο κύριος Πρέντα για την Ισλανδία. Ρέντα, θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην 6 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στο 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά,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 αποχές εγκρίνεται προφορική έλεγχος. Die Liberalen haben diesmal zugestimmt. Ψήφισαν υπέρ αυτή τη φορά. Πέρα ψηφοφορία. 35 υπέρ, 27 κατά, εγκρίνεται. Τώρα προφορική τροπολογία 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική 6 υπέρ. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Πάντα με προφορική τροπολογία λέει ο πρόεδρος. The Green Group, unfortunately, is totally... Η πράσινη, η ομάδα μας, αντιτασσόμαστε στις προφορικές, σε οποιαδήποτε προφορική. Μάλιστα, τότε ψηφίζουμε μόνο την συμβαστική 6 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής 6 χωρίς την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 38 υπέρ. Κατά. αποχέ. Τι έκανε οι χειριστέ πώς ψήφισαν. Έλεγχος, έλεγχος, ε, έλεγχος. 38. 38. Yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρα ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Η 39, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ. Καταπίπτει, καταπίπτει, λόγω της 38. Συμβαστική 7, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 3. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Yeah, the closed vote is closed. Πέρα ψηφοφορία, 56 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Πέντε λεπτά. President, Ambassadors, friends, I would like to welcome... Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, τον κύριο Ράνκο Κρυβοκάπιτς. Χαίρομαι που είστε μαζί μας σήμερα και νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνονται οι συζητήσεις αυτές. Το 2006 ήρθατε εδώ πέρα στην Επιτροπή τη δική μας πριν από την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος σε μια σημαντική ε, χρονική στιγμή. Θα θυμάστε και εμείς θυμόμαστε ασφαλώς το τι συνέβη έκτοτε δεν θα ήταν εύκολο για τους αντιπαλούς σας. Το τελευταίο μήνα υιοθετήσαμε συστάσεις ε, για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Θεωρούμε από πολλές απόψεις ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί θετικό παράδειγμα στην περιφέρεια και είναι μάλιστα η μοναδική χώρα στην περιφέρεια που βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης ε, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι υποδειγματική η εξέλιξη και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών του Μαυροβουνίου. Για να αναφέρω έτσι ενδεικτικά κάποια επιτεύγματα για τα οποία μπορεί να περηφανευτεί η χώρα σας. Τα επιτεύγματα αυτά φυσικά θα πρέπει να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν για την ευημερία των πολιτών όλης της περιφέρειας και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνοντας ε, την δικαστική ανεξαρτησία, την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, την ε, συνεργασία σε περιπτώσεις εγκλήματος αύξησης της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους γείτονές σας. Σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος που θα λάβετε το λόγο. Αλλά θα ήθελα καταρχάς να καλέσω τον συνάδελφο Κούκα να κάνει κάποια σχόλια. Πρωτού κύριε Πρόεδρε λάβετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οποία τιμή να λαμβάνω το λόγο πριν τον πρόεδρο της Μαυροβουνικής Βουλής. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο, τον κύριο Κρυβοκάπιτς, στην Επιτροπή μας και από την εμπειρία που είχαμε από την διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία μπορώ να επιβεβαιώσω ότι στις συζητήσεις με τους συνομιλητές μας από το Μαυροβούνιο μπορούμε και εμείς να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι συνομιλητές μας αντιμετωπίζουν με πολύ υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τις περίπλοκες και επίμεχες μερικές φορές τις καταλήγουμε πάντα σε υιοθέτηση κοινή δήλωσης. Η πολιτική του Μαυροβουνίου και η παιδεία πολιτικού διαλόγου υπάρχει στο Μαυροβούνιο. και ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενθαρρύνω κύριε Πρόεδρε να συνεχίσετε τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις με τον ίδιο ρυθμό και θα ήθελα να τονίσω και εγώ αυτό που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται σε προενταξιακές διαπραγματεύσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη δυναμική της διεύρυνσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και είναι ευχής έργων που συνεχίζει τη διαδικασία αυτή το Μαυροβούνιο και θα πρέπει να επενέσουμε τη χώρα αυτή ε, βέβαια, το γεγονό ότι είναι η μοναδική χώρα τη περιοχή που συνεχίζει πρωταξιακέ διαδικασίε ε, φέρει στου ώμου του τεράστια ευθύνη. Γιατί χρειαζόμαστε κάποια παραδείγματα από τι χώρε των Βαλκανίων ότι είναι δυνατή η ένταξη, όπω συμβαίνει με την Κροατία. Εφόσον οι υποψήφιε χώρε εκπληρώνουν τι υποχρεώσει του και τι προποθέσει για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εφικτή η προσχώρησή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το επιχείρημα γιατί πολλοί μας κατηγορούν ότι οι Ευρωπαίοι δεν κρατάνε το λόγο τους και δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Όχι όμως, μπορούμε να το διαψεύσουμε αυτό. Δεν έχω κανένα αρνητικό σχόλιο και γνωρίζετε ε, θαυμάσα τα προβλήματα, είστε πολύ εξοικειωμένοι και γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκκρεμή προβλήματα. Ευτυχώς που ξεκινάνε ξεκίνηση διαπραγματεύσεις με τα κεφάλαια 23 και 24, γιατί είναι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα σε πολλές χώρες αυτά τα δύο κεφάλαια. Πάντως αυτή η διαπραγματευτική μέθοδος είναι πολύ πιο αποτελεσματική, γιατί μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο επίμαχα, καθόδια, αλλά και τα πιο σημαντικά ταυτόχρονα ζητήματα. Ευχαριστώ. Thanks a lot, Mr. President Brock. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπροκ. Λίγους μήνες πριν από την ανεξαρτησία εξηγήσαμε εδώ πόσο σημαντικό ήταν ε, για εμάς να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρώπη. Χαίρομαι γιατί τα καταφέραμε πολύ καλά κατά τον σωστό τρόπο και δείξαμε στις υπόλοιπες βαλκανικές ε, χώρες πόσο ε, τα δύσκολα ζητήματα μπορούν να επιληθούν ε, ειρηνικά και παραγωγικά. Συναντήθηκα με τέσσερις προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ένας βρίσκεται εδώ μεταξύ μας, ο κύριος Πέτεριν, και κάθε φορά ε, με κατακλείς μεγάλη χαρά να τους συναντώ, να σας συναντώ. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να τον ευχαριστήσω και προσωπικά τον κύριο Πέτερινγκ Έχουμε μεταξύ μας και τον Αντιπρόεδρο Κούκαν μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Σταθερότητας και ε, Σύνδεσης και εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε τέσσερις φορές το χρόνο, ιδιαίτερα στα κεφάλαια 23 και 24 που είναι τα βασικά κεφάλαια για το Μαυροβούνιο. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τα νέα στοιχεία που διέπουν τις σχέσεις μας. Ε, προσωπώ το νέο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου και φυσικά το κοινοβούλιο, το μεγάλο κοινοβούλιο είναι το, το σημείο διεπαφής και ένας βασικός θεσμός ένωσης, ενωτικό στοιχείο για το Μαυροβούνιο, αν και πολλοί είχαν ταχθεί κατά της ένταξης. Τώρα το Κοινοβούλιο εργάζεται στεναρά για να αλλάξει το Σύνταγμα, Παλά το γεγονός ότι ε, αλλάξαμε, μεταρρυθμίσαμε το Σύνταγμα το 2007, δηλαδή ένα χρόνο μετά την ανεξαρτησία. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και το διοδοτικό, συγχωρείτε, σύστημα, το δικαστικό κλάδο και να ορίσουμε ένα σταθερό πλαίσιο για την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου αλλά και τη λογοδοσία του. Δεν πρόκειται για μια ανεξάρτητη εξουσία η οποία δεν φέρει μεγάλες ευθύνες, φέρει μεγάλες ευθύνες και είναι υπεύθυνη για ε, γενικότερα θέματα νομιμότητας. Εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε το σύνταγμά μας και να προωθήσουμε την ανεξαρτησία αλλά και τη λογοδοσία του δικαιοδοτικού τομέα. Ελπίζω ότι το νέο κοινοβούλιο μέσα στο πλαίσιο της, ε, των συνταγματικών αλλαγών θα το επιτύχει τους επόμενους ε, μήνες. Το Μαυροβούνιο θα αποδείξει πώς μπορεί τάχιστα να αλλάξει τα πρότυπα που διέπουν το δικαιοδοτικό τομέα, όπως είδαμε και στα κεφάλαια 23 και 24. Έχουμε υψηλές προσδοκίες. Επίσης υπάρχει πραγματικός έλεγχος του εκτελεστικού. Έχουμε, είχαμε 26 ακροάσεις στο Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου και αυτό που είναι μοναδικό στην κοινοβουλευτική μας ζωή είναι ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, 15 μέρες πριν από τις εκλογές, ο επικεφαλής ε, ενός βασικού κόμματος και τώρα ο πρωθυπουργός, ο νυν υπήρξε άμεσα ενδιαφερόμενος και έτυχε και έρευνας, δηλαδή διερευνήθηκε περίπτωσή του πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Και αυτό δείχνει, καταδεικνύει το, την κοινοβουλευτική δημοκρατία της νέας αυτής χώρας. Ελπίζω στο εγγύς μέλλον να συνεχίσουμε με αυτές τις δραστηριότητες Επίσης υπάρχουν πάχνες ακροάσεις για την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, την Επιτροπή Ασφάλειας και οι βασικές ε, επιτροπές για τον προϋπολογισμό, για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται στα χέρια της αντιπολίτευσης. Ξέρετε ότι η Επιτροπή του προϋπολογισμού είναι ύψης της σημασίας, αλλά αυτό αφορά και την Επιτροπή κατά της ε, διαφθοράς και την Επιτροπή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα καθήκοντα ένταξης, τα καθήκοντα προσχώρησης και στη διαδικασία ελέγχου έχουμε εντάξει και τον τομέα των ΜΚΟ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η κοινωνία ε, κινητοποιείται γενικότερα και έτσι όλα, ολόκληρος ο κοινωνικός ιστός ασχολείται με θέματα ενταξιακά, καθαρά θέματα ένταξης, για να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις και για την εφαρμογή των αξιών της Ευρώπης. Επιπροσθέτως θα ήθελα να πω ότι την επόμενη φορά που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι πιο ε, ε, αποτελεσματικά δυνάμει των κεφαλαίων 23 και 24. Και αυτό αφορά όλες τις κοινωνίες, όχι μόνο τις ε, νέες δημοκρατίες, δηλαδή να δώσουμε πραγματικό νόημα στο κράτος δικαίου. Έχει μεγάλη σημασία για όλες τις κοινωνίες και είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ε, σημάδι μίας όριμης κοινωνίας. Ελπίζω λοιπόν κατά τη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου να ανταποκριθούμε σε όλα τα επίπεδα γιατί έχει σημασία η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων σε όλους αυτούς τους τομείς. Και αυτό που έχει σημασία... Για το τέλος ομιλίες, γιατί βλέπετε τελειώνει ο χρόνος μου το, Μαυ... Μαυροβόνιο που είναι μια μικρή χώρα είναι ένα καλό υπόδειγμα πολυεθνοτικής κοινωνίας γιατί και πολυπολιτισμικής. Έχουμε στη χώρα μας, στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί. Είμαστε το σταυροδρόμι πολλών ιστορικών πολιτισμών και η παράδοση στην κοινωνία μας είναι ότι μια πολιτιστική, πολυπολιτισμική και πολυεθνωτική κοινωνία είναι σημαντική και πλούτος. Και αυτό, ήταν, αυτό ε, είναι μια παράδοση που την έχουμε από το παρελθόν, από τη Βασιλεία. Ο Βασιλιά ήταν αρκετά έξυπνο ώστε να θέλει να εντάξει όλε τι διάφορε εθνότητε και πολιτισμού ε, στο Μαυροβούνιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω γιατί όλου μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια κοινωνιακή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινωνία που είναι ανταγωνιστική προς τις υπόλοιπες του κόσμου, αλλά θέλουμε να δώσουμε ένα σωστό παράδειγμα, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση για την περιοχή και να βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση ε, της ε, περιοχής αυτής, σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης ε, που θα στηρίζεται σε, στη Βουλή Ανεξάρτητων Χωρών. Περάσαμε πολλά, ειδικά στη δεκαετία του 1990. Είχαμε όμως πολύ θετική κληρονομιά και πολλά επιτεύγματα και κατορθώματα τους τελευταίους αιώνες. Πιστεύω ότι μπορούμε να επαναντάξουμε ε, τα Βαλκάνια με μια νέα βάση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ και 10 χρόνια έχουμε συστήσει ένα διακοινοβουλευτικό φόρουμ. Και μάλιστα ήταν μια πρώτη πρωτοβουλία των Δυτικών Βαλκανίων Εκεί προσπαθούμε να επανασυμφιλιώσουμε τα διάφορα κράτη της περιοχής και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με όλα τα τοπικά κοινοβούλια, τα κοινοβούλια των γειτονικών χωρών. Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί σταθήκατε από την αρχή στο πλευρό μας. Μόλις ε, ολοκλήρωσε την επίσκεψή της Doris Πακ και ο Τσαρλ Στάνοκ ε, μας βοήθησε πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ επίσης είναι στο πλευρό μας μαζί με όλους τους άλλους. Ξέρουμε ότι έχουμε φίλους ε, εδώ στην Ομίγυρη και οι φίλοι δείχνουν κατανόηση όταν κάνει κανείς ε, λάθη αλλά βοηθούν, τον βοηθούν και να τα διορθώσει. Και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που δείξατε στο Μαυροβούνιο και θα ήθελα να εκφράσω την ευτυχία μου γιατί βλέπω ότι ε, έχουμε πολλούς παρατηρητές από την Κροατία στην Επιτροπή αυτή και όσον όπου η Κροατία θα γίνει πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μας είναι αυτό μεγάλη ενθάρρυνση και δίνει πολλά ενάυσματα και ελπίζω ότι και εμείς στο μέλλον θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Ευχαριστώ. President, Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά για την εισαγωγή. Πρώτα ζήτησε το λόγο ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον πρόεδρο της Μαυροβουνικής Βουλής. λοιπόν, που δεν ήμουν από την αρχή της συνεδρίασης για να ακούσω την ε, ομιλία σας. Αλλά ξέρετε ότι η έκθεσή μου πέρασε στο Κοινοβούλιο ε, σχεδόν πανψηφή. Ε, βέβαια, συντάχθηκαν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως πιστεύω ότι η τελική μορφή της έκθεσης είναι πολύ ικανοποιητική. Και εγώ ως φίλος του Μαυροβουνίου γνωρίζω ότι είναι καλή η επικοδομητική κριτική και αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα τη σωστή πορεία της χώρας σας παρά τις ε, επικρίσεις που μπορεί να έχουμε ασκήσει καλοπροαίρετα πολλές φορές και τα κεφάλαια 23 και 24 και το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος της διαφθοράς βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του προγράμματος των διαπραγματεύσεων, είναι ύψη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα σημεία αυτά ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάλια. Πάντως είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να εκπληρώσει προϋποθέσεις, ε, για να ανοίξει και να κλείσει αισίως τα κεφάλαια αυτά. Ξέρω ότι ε, το, το ζωηρό το ενδιαφέρον που ξύπνησε η έκθεση, υποβλήθηκαν πολλές τροπολογίες για τα θέματα των μειονοτήτων, περιβάλλοντος, εσωτερικά εκτοπισμένους, ε, και σίγουρα για μια μικρή χώρα έχετε διανύσει τεράστιο δρόμο και βελτιώσετε το θέμα της παρακολούθησης και νομίζω ότι υπάρχει πια μεγάλη συνένεση ε, στο Μαυροβούνιο υπέρ της ε, ενταξιακής πορείας. Και ε, η χώρα είναι μικρή, δεν ταλανίστε από τέτοια προβλήματα που έχουν κάποιοι γειτονές σας και ελπίζω το εκρεμές, η εκρεμής διαφορά για τα σύνορα με την Κροατία δεν θα α, σας προβληματίσει διμερώς για πολύ ακόμη καιρό και ελπίζω ότι με το που θα μπει Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιληθεί το πρόβλημα και ελπίζω να διαμεσολαβήσετε ώστε να εκτονωθούν οι εντάσεις που υπάρχουν και σε γειτονικέ χώρες όπως η Ελβανία η Βοσνία, η και άλλες. Πάντως αυτή τη στιγμή εσείς πρωτοστατείτε στα Δυτικά Βαλκάνια ε, στα πλαίσια της ενταξιακής διαδικασίας και θα σας παρακολουθεί εκ του σύναγκης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο όσο προχωρείτε σε αυτή την ενταξιακή σας πορεία και στην πορεία σας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτά ευχαριστώ. Thank you. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε αναφέρετε τους φίλους σας. Έχετε πολλούς φίλους εδώ στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο ε, εδώ στην Επιτροπή και φυσικά οι σοσιαλδημοκράτες είμαστε φίλοι σας και προωθούμε την ε, ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθούμε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με όλες τις χώρες της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου και του Μαυροβουνίου. Φυσικά, εσείς θα πρέπει να κάνετε τα μαθήματά σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί φυσικά εμείς μπορούμε να σας ενθαρρύνουμε, να σας υποστηρίξουμε, αλλά εσείς θα πρέπει να κάνετε τα μαθήματά σας. Ενθαρρυντικό το ότι ακούσαμε λοιπόν ότι υπάρχει ομοφωνία στο Μαυροβούνιο, γιατί αυτό αποτελεί τη βάση. Είναι καλό ότι υπάρχει ομοφωνία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των κομμάτων. Είναι θετικό αυτό. Το ότι το ακούμε αυτό, αυτό από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά τους προέδρου των επιτροπών κτλ. Αλλά και σε ό,τι αφορά και την ε, αντιπολίτευση. Φυσικά γνωρίζετε τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς μέχρι τη λειτουργία του κράτους, ε, της κυβέρνησης, της διοίκησης. Ξέρετε νομίζω τι έχετε να κάνετε και βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Επίσης, αυτό που είναι ε, εξίσου σημαντικό και αυτό που καλούμε και αποκαλούμε εμπειρία των νέων κρατών μελών, είναι σημαντικό μια χώρα να προετοιμάζεται όχι μόνο σε διοικητικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί όταν θα ενταχθείτε σε αυτή τη μεγάλη αγορά 500 εκατομμυρίων ατόμων και καταναλωτών, αυτό θα δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες, αλλά και κάποια πίεση στη δική σας οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πώς θεωρείτε ότι εξελίσσεται και αναπτύσσεται η οικονομία σας, γιατί δυστυχώς ζούμε σε εποχές όπου οι περισσότερες, αν όχι όλες οι χώρες μας, νιώθουν τον αντίκτυπο της κρίσης. Ε, φυσικά υπάρχει αντίκτυπος και στη δική σας χώρα. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα κονδύλια, τα πρωτεντεξιακά, αλλά σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη ενοποίηση ήδη των οικονομιών μας πριν ενταχθείτε στην Ένωση. Τελευταία παρατήρηση αναφέρθηκε ήδη ότι το Μαυροβούνιο είναι στην ε, κορυφή αν θέλετε και η Κροατία είναι πριν από εσά. Θα ενταχθεί η Κροατία από 1η Ιουλίου και μετά θα είναι η δική σας σειρά. Αυτό σημαίνει και μια μεγάλη ευθύνη γιατί εσείς ανοίγετε το δρόμο για τους φίλου στην ε, Αλβανία, στη Βοσνία, στη Σερβία. Εσείς καταδεικνύετε ότι όταν δουλέψει κανείς σκληρά μπορεί να πετύχει. Το αναφέρατε. Ξέρετε ότι το, το Μαυροβούνιο θα διαδραματίσει αυτό το σημαντικό ρόλο όχι μόνο για το εσωτερικό της χώρας, αλλά και για όλη την περιφέρεια και για όλες τις μελλοντικέ διευρύνσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Κύριε Μπρισάτζιτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε στο δικό μας κοινοβούλιο κύριε Πρόεδρε της Βουλής. Όπως ε, είπα και συνάδελφοι, η χώρα σας ήταν μια πολύ ε, πετυχημένη περίπτωση. Και όλοι η Ρεν ήταν επίτροπος που είπε πριν από 7-8 χρόνια ότι ε, ήσασταν επιτυχημένη ιστορία. Έχουν περάσει 8 χρόνια και εξακολουθούμε να σας αποκαλούμε ως πετυχημένη εμπειρία. Είστε μια από τις μικρότερες χώρες ε, στην περιοχή, αλλά με τις μεγαλύτερες ε, φιλοδοξίες θα έλεγα. Και εξακολουθείτε την επιτυχημένη σας πορεία. Εγώ πιστεύω ειλικρινά, γι' αυτό και πίεσα να ξεκινήσουν οι ε, διαπραγματεύσει ενταξιακέ με το Μαυροβούλιο, γιατί πιστεύω ότι μόνο όταν ξεκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει ε, θα δοθούν τα ενάψματα για τι σωστέ μεταρρυθμίσει. Τώρα, ε, ω χώρα που διαπραγματεύεστε για την ευρωπαϊκή, για την ευρωπαϊκή ένταξη, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι με το που πραγματοποιείτε ένα βήμα θα πρέπει να είστε έτοιμοι για το επόμενο. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μιας χώρας σαν τη δική σας και τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, που ίσως δεν πιστεύουν ακόμη στις μεταρρυθμίσεις, γιατί δεν είναι σίγουροι για το μέλλον τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να σας, να σας κάνουμε κήρυγμα και να σας δίνουμε μαθήματα, αλλά να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο κινητήριος μοχλός των μεταρρυθμίσεων είναι να δοθεί μια ρεαλιστική και εφικτή προοπτική για τις διαπραγματεύσεις. Όταν μια χώρα γνωρίζει ότι ναι, δεν θα χρειαστεί να κάνει μεταρρυθμίσεις, αλλά θα έχει μια επιβράβευση ε, και μια πρόοδο στην ενταξιακή της πορεία θα έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο για να τις πραγματοποιήσει. Το ξέρετε και εσείς καλά, ξέρετε ότι θα πρέπει να εντείνετε τις προσπάθειές σας. Εγώ μπορεί να μην είμαι τόσο δραστήρια όσο ο κύριος Στάνο, γιατί είμαι μια πλησκιώδη συγγήτρια για την έκθεση Τάνοκ, αλλά δεν κατέθεσα καμία τροπολογία στην έκθεση Τάνοκ, γιατί θεωρώ ότι ήταν πολύ εύστοχη και για τις θετικές πτυχές της διαπραγματεύτική διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα και επισήμανε τα κενά η έκθεση του κυρίου Τάνοκ. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι είστε μια πολύ επιτυχημένη χώρα και γι' αυτό δεν ήθελα να υποβάλλω πολλές τροπολογίες, γιατί και εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ο ρόλος σας στην περιοχή ήταν πραγματικά ηγετικός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον για θέματα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Τώρα, με την έναρξη των ανταξιακών διαπραγματεύσεων θεωρείτε ότι τα θέματα συνεργασίας και καλής γειτονίας θα παραμείνουν προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας. Γιατί μια, για μια χώρα που δεν είχε αναμειχθεί και πολύ ενεργά σε θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα για τα Βαλκάνια. Εσείς δεν ε, κάνατε πολιτικές επεμβάσεις, στρατιωτικές επεμβάσεις, συγγνώμη, σε γειτονικέ χώρες. Είστε από τις λίγες χώρες που όταν οργανώνετε συνεδριάσεις ε, έρχονται όλοι προσκεκλημένοι, δεν σας μποϊκοτάρει κανένας. Είστε από τις λίγες χώρες που έχει τέτοια πολυτέλεια και αυτό μπορεί να διαδραματιστεί ηγετικό ρόλο σε θέματα περιφερειακών σχέσεων και περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ελπίζω βέβαια να μην αποσπαστεί η προσοχή σας και να μην επικεντρωθεί μόνο στην ε, ενταξιακή διαδικασία. Κυρία Πάκ, σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε και να πω και στον κύριο Ρούτσεκ ότι δεν χρειάζεται να ζηλεύει γιατί δεν ανήκει στη δική μου οικογένεια αλλά έχουμε την πολιτική οικογένεια, αλλά είμαστε φίλοι εδώ και 20 χρόνια, άρα δεν χρειάζεται, χρειάζεται να ζηλεύεις σίγουρα προς τη δική σου ε, πολιτική οικογένεια. Τι είναι παρά προς τη δική μου. Παρ' όλα αυτά, ε, τον συμπαθώ ιδιαίτερα και μπορούμε να του λέμε τι δεν μας αρέσει. Και αυτό είναι το καλό με το Μαυροβούνιο, ότι μπορούμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό είναι πλεονέκτημα, αυτό που είπε και η συνάδελφος ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μευροβούνιο δεν είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι γειτονικέ του χώρε. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα σε σχέση με τι γειτονικέ χώρε όπου υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε αυθεντικέ ε, εντάσει. <coughs> Πε μα, τι... τι γίνεται με τις μειονότητες, με την αλβανική, με τη βοσνιακή μειονότητα και με το μεγάλο ποσοστό των Σέρβων που υπάρχουν ακόμα. Έχετε προβλήματα, θα μπορούσατε να μας πει δύο λόγια και να τονίσω αυτό που είπε και η Άννα. Να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το φόρουμ για την περιφέρεια. Θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται δίνουν τη δυνατότητα στον ε, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να προωθήσει αυτή την διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης και νομίζω ότι αν μας καλέσετε ε, ασφαλώς και θα είμαστε και εμείς ε, διατεθειμένοι να μεταβούμε για να σας βοηθήσουμε στις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εξ ονόματος των ε, Πρασίνων θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο κοινοβούλιο μας. Είναι πολύ θετικό το ότι βρίσκεστε εδώ για να συζητήσουμε ε, ανάμεσα στις επίσημες ε, συναντήσεις που προβλέπονται. Επίσης, δέχομαι με χαρά το γεγονός ότι είπατε ότι το κοινοβούλιο σας είναι ένας ενωσιακός, ενωτικός παράγων όταν μιλάμε για την ενταξιακή διαδικασία και η ε, Doris Πάκ σας ε, μίλησε για τις ε, σχέσεις μεταξύ Σέρβων και Μαυροβουνίων Μπορείτε να μας πείτε πώς εξελίσσονται τα πράγματα ως προς τις διμερείς σχέσεις. Υπήρχαν προβλήματα ως προς τον εθνικό ύμνο, τη σημαία και ούτω καθεξής. Ξέρετε ότι είμαι φίλη του Μαυροβουνίου, αλλά θα πρέπει να είμαι και επικριτική το γεγονός ότι τώρα διαπραγματευόσαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι έχουν ανοίξει τα κεφάλαια 23 και 24 είναι κάτι το θετικό όχι μόνο για το Μαυροβούνιο αλλά για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί μετά την Κροατία είσαστε η αμέσως επόμενη χώρα όπου δεν υπάρχουν προσκόμματα, τόσα πολλά προσκόμματα όσα αναμένονταν. Επίσης έγινε λόγος για την ελευθερία τύπου. Ε, είχαν ακουστεί απειλές κατά των δημοσιογράφων. Πολλοί προσήχθησαν στα δικαστήρια, οι πέτοι, αλλά η αδελφή του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή έχει κάνει μήνυση σε δύο ε, εφημερίδες και δημοσιογράφους μέσα στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης της Telecom είναι κρίσιμο το θέμα και τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχουν επιληφθεί του ζητήματος, αλλά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Επίσης δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος σε περίπτωση άλλων απειλών κατά δημοσιογράφων. Πολλοί δημοσιογράφοι φοβούνται ότι επειδή είναι επικριτικοί έναντι της κυβέρνησης, υφίστανται πιέσεις και θα λάβουν οι επιχειρήσεις τους λιγότερες διαφημίσεις, δεν θα έχουν τόσο διαφημιστικό ε, χρόνο ή χώρο. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα, το γνωρίζω, αλλά σας επισύρω την προσοχή σε αυτό ως προς την ε, ελευθερία των ε, ΜΜΕ. Επίσης η εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο σας είναι ένα θέμα ήταν ένα θέμα. Μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας μιλήσατε για συμμετοχή ενός 30% γυναικών. Η εκπροσώπηση ανέρχεται σε 17% των γυναικών. Εσείς ως πρόεδρος της Βουλής τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να φτάσετε στο ποσοστό το 30% ε, εκπροσώπησης των γυναικών. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πολύ καλή η εκπροσώπηση. Δηλαδή, τη στιγμή που το υποσχεθήκατε προεκλογικά, καλό θα ήταν και να ανταποκριθείτε, δηλαδή να, να τηρήσετε, να κρατήσετε το λόγο σας και να μην αφήσετε τις γυναίκες πίσω. Και κάτι άλλο. Το Μαυροβούνιο είναι ε, πολύ μπροστά στα Δυτικά Βαλκάνια ως προς την εκπροσώπηση λεσβιών, ομοφιλοφίλων κλπ. Η προηγούμενη κυβέρνηση ζήτησε ε, από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης να ανταποκριθούν στη σωστή εκπροσώπηση, στη σωστή αντιμετώπιση του θέματος. Δεν χρειάζεται να σας προτρέπουμε εμείς πάντα για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να μας πείτε πώς το Κοινοβούλιο θα δραστηριοποιηθεί και σε αυτό το τομέα. Ε, προσμένω σε μια πολύ καλή και αγαστή συνεργασία και στο μέλλον. Thank you, Chair. Ο κύριος κύριε Πρόεδρε, καλώς και εκ μέρους των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγχαρητήρια για όσα έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Και ελπίζω ότι στη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας θα ρίξετε και πολλά νέα κεφάλαια. Γιατί αυτό περιμένουμε απεγνωσμένα από εσά και αυτή θα είναι, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό κίνητρο για τους Ντάτσιτς και Θάτσι που βρίσκονται στις Βρυξέλλες προκειμένου να καταλήξουν σε ίσως ιστορική σημασία συμβιβασμό και θα είναι και ένα σημαντικό μήνυμα στις υπόλοιπε χώρες της περιοχής γιατί ε, από τη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο σίγουρα το Μαυροβούνιο έχει τις καλύτερες επιδόσεις είναι ε, παράδειγμα προς μίμηση. Ενώ άλλες ε, χώρες της περιοχής δυστυχώς είναι κάπου χαμένες ε, στην ιστορία και δεν ε, ατενίζουν το μέλλον, αλλά κάπου έχουν μπλοκαριστεί στο παρελθόν. παρά τις δηλώσεις που έγιναν για το μέλλον του Μοντενέγκρο, ένα, μία από τις δηλώσεις ήταν να, να επιληθεί το θέμα των ΛΟΑΔ, λεσβιών, ομοφιλοφίλων, φιλομεταβατικών κλπ. και να μην ε, ε, γίνουν κάποιες μυσαλόδοξες δηλώσεις ή ε, μια έξαψη των, του μίσους. Κατά τη γνώμη μου τέτοιες μυσαλόδοξες δηλώσεις είναι εξωπραγματικές, για να μην πω εξωγήινες. Εγώ θεωρώ ότι το Μαυροβούλιο θα πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερο προκειμένου να αναπτύξει το διάλογο μεταξύ όλων των κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και της κυβέρνησης για τα θέματα αυτά. Αυτό που έγινε και υπόθηκε φαίνεται αγνώρισε και εμένα τέτοιου είδους μηνύματα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για στρατηγική ή για τακτική. Αλλά αν πρόκειται για τακτική, πραγματικά είναι πολύ λάθο αυτή η για τακτικη αλλα αν προκειται για τακτικη πραγματικα ειναι πολυ λαθος αυτη η τακτικη Θεωρώ ότι το σύστημα των αξιών ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει σταδιακά να εφαρμοστεί και στο Μαυροβούνιο και όχι μόνο α, ε, όπως είπε η Ούλρικε σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά σε κάθε διάλογο που έχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή εκπρόσωποι τους με την κυβέρνηση η κυβέρνηση, αν θεωρεί, ή με την Εκκλησία, θεωρήσουμε ότι η Εκκλησία μπορεί να θεωρηθεί με κυβερνητική οργάνωση. Thanks uh, Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ναι, η οικονομία, όπως ε, και όλοι οι υπόλοιποι, πληρώνουμε τώρα το τίμημα κατά κάποιο τρόπο της ε, φούσκας των ακινήτων. Η Βουλγαρία, η Ισπανία, και όλοι οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε, είμαστε μικρή επικράτεια. Έχουμε πολλές επενδύσεις στις υποδομές, στην ενέργεια. 20% χρησιμοποιούμε ε, από υδροελεκτρικές πηγές ενέργειας και θερμική ενέργεια. Θα συνεχίσει η ανάπτυξη. Βρισκόμαστε στο 0,5% ε, σε επίπεδα ποσοστά ανάπτυξης. Ε, υπάρχει δυναμικό αν δεν χάσουμε τουλάχιστον ευκαιρίε όπω την προηγούμενη φορά, θα είμαι, είμαι αισιόδοξο για το οικονομικό μέλλον μα. Συζητούσα με τον Πρωθυπουργό Μιλάνο τη Κροατία. παλιό μου φίλο, για τουριστικές προσφορές και από πολιτικής άποψης πρέπει να πω ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες στο Μαυροβούνιο και να τονώσουμε τις σχέσεις με την Κροατία. Άννα, σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη. Δεν σε ανέφερα, αλλά ασφαλώς και μας υποστηρίζετε σε ό,τι αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός. Πρέπει να πω ότι Έχω 24 χρόνια περάσει στο κοινοβούλιο, σε κοινοβούλια τεσσάρων χωρών και έχω εμπειρία από τα κοινοβούλια. Το Μαυροβούνιο αποτελεί τον πυρήνα της σταθερότητας και της ισορροπίας στην περιφέρεια. Μιλάμε για ισορροπία, όχι μόνο για σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ μικρή χώρα, αλλά με πολύ θετικό αντίκτυπο στην σταθερότητα στην περιοχή και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη θέση αυτή, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις εκείνες, ιδιαίτερα στην κοινωνική ζωή. Η Ντόρις ανέφερε κάποια παραδείγματα για να βελτιώσουμε, για παράδειγμα, τις δυνατότητες του φόρουμ και να βελτιώσουμε και τις ε, συνεργασίες μεταξύ των κοινοβουλίων, με τους ε, συναδέλφους μεταξύ της Κροατίας, της Μακεδονίας, λέμε της. Και το κοσυφοπαίδιο. Αυτό θα γίνει και στο μέλλον όπως το έχουμε κάνει και ιστορικά, στον 19ο αιώνα. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να συνενώνουμε τις ε, τάσεις από την Κροατία, από τη Σερβία. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό για το Μαυροβούνιο και πολλοί από τους ε, οι ηγέτε μα χρησιμοποίησαν αυτέ τι ιδιότητε σε διάφορε ιστορικές ε, στιγμέ. Αναφέρθηκα στο φόρουμ να αναφερθώ στις μειονότητε. Ξέρετε ότι έχουμε κάποιε ιδιαίτερε μειονότητε, μη τυπικέ στο Μαυροβούνιο. Οι τυπικέ μειονότητες είναι οι Αλβανοί και είναι δεσμευμένοι, υποστηρίζουν πάρα πολύ το κράτο του Μαυροβουνίου. Πιο πολύ από ότι η ορθόδοξη ε, πλειοψηφία, πλειονότητα. Αυτό δεν είναι τυπικό βάση της ε, ιστορίας μας. Ο βασιλιάς μας ε, ε, μεταχειρίστηκε διαφορετικά τις Ισλαμικές ε, μειονότητες. Τους άφησε τις ε, στρατιωτικές μονάδες, το, τη Σαρία για 10 χρόνια. Το Μαυροβούνιο, μην ξεχνάτε ότι το 19ο αιώνα χαρακτηρίζεται από θεοκρατία, χριστιανική θεοκρατία μέχρι το 1851. Αλλά αυτή η οριμότητα έχει θέσει τις βάσεις για την κοινωνία του 21ου αιώνα. Υπάρχει εμπιστοσύνη γιατί υπήρχε αυτή η βάση από τον 19ο αιώνα. Δεν θέλω να πω και να μιλήσω για τη σερβική μειονότητα ένα σαρδικό έθνος στο Μαυροβόνιο. Όπως όλες οι υπόλοιπες ε, εθνότητες. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ το, τον όρο μειονότητα. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, γιατί είναι μεγάλη η παράδοση. 9% Σέρβοι στο 91 και τώρα 27% Σέρβοι. Μιλάμε πιο πολύ για πολιτική έκφραση και όχι τόσο για εθνοτική έκφραση. Τι κάναμε λοιπόν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Σέρβος από τη Νέα Σερβική Δημοκρατία. Ήταν κατά της ανεξαρτησίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κατά της διαφθοράς ήταν ο ηγέτης του κινήματος για την Ένωση με την Σερβία. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών ήταν εκείνος που ήταν κατά της ανεξαρτησίας. Έτσι λοιπόν ενσωματώνονται και προσπαθούμε να βάλουμε τις ε, διαφωνίες μας στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ούτω καθεξής. Έτσι, έτσι ενοποιούμαστε, ενσωματώνουμε όλα τα άτομα και τις ρίζες μας στο Μαυροβούνιο, γιατί βλέπετε στο Μαυροβούνιο ε, ακόμα και η Δερφείο. ο ένας είναι Σέρβος και ο άλλος είναι Μαυροβούνιος. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η βάση για την αισιοδοξία για τους νέους μαυροβούνιους έχουν διαφορετικές θρησκείες, είναι μουσουλμάνοι, ορθόδοξοι, χριστιανοί. Εκφράζονται ως μαυροβούνιοι παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικές ρίζες. Αυτό τι σημαίνει ότι αναπτυσσόμαστε, αναπτυσσόμαστε όχι ως εθνικό κράτος. Ποια είναι η βάση στο σύνταγμά μας, δεν είμαστε το κράτος ε, των Μαυροβούνιων, είναι των Είμαστε κράτο των πολιτών του Μαυροβουνίου και αυτό έχει σημασία για το μέλλον του Μαυροβουνίου, για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Οι δύο πιο έγκυρε ε, εφημερίδες που πουλούν πιο πολλά αντίτυπα στο Μαυροβούνιο είναι τη αντιπολίτευσης. Η μία εξ αυτών έχει ουσιαστικά δημιουργήσει το κόμμα, η άλλη υποστηρίζει τα κόμματα υπέρ της Σερβίας. Υπάρχει ελευθερία, ακόμα και αν δεν υποστηρίζει κανείς την κυβέρνηση. Και ναι, για τις υποθέσεις που αναφέρατε χρειάστηκε να τις επιλύσουμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια ισορροπία δυνάμεων με τη Σερβία. Έχουμε και την καταγγελία της αδερφής του Πρωθυπουργού κατά της εφημερίδας. Ας μην, μην ξεχνάμε όμως η Deutsche ε, Telekom εξετάστηκε από Επιτροπή του Κοινοβουλίου και η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να ζητήσει α, διεξαγωγή έρευνας. Δεν προστατεύθηκε. Έχει καθήκον να προσέλθει στο Κοινοβούλιο και να λογοδοτήσει αν κάποιος το ζητήσει. και να μην ξεχνάτε ότι το κάναμε αυτό κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της προεκλογικής για τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές. Έτσι προσπαθούμε να πετύχουμε μια ισορροπία. Ξέρετε ότι αποποινικοποιήσαμε τις, τα σχόλια, τη δυσφήμιση. Δεν περιλαμβάνεται πλέον στο ποινικό μας δίκαιο, δεν προβλέπεται. Και θεωρώ ότι προχωρούμε προς τα εμπρός στον τομέα αυτό εκο, για την Σερβική Εκκλησία στο Μεσοβούνιο. Ο Πρωθυπουργό και εγώ έχουμε το ίδιο θέμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεωρώ ότι πολύ μεγάλο τμήμα τη ε, προεκλογική του εκστρατεία συνδέεται με αυτό, όχι τόσο πολύ με το οργανωμένο έγκλημα, παρά το γεγονό ότι στην πολιτική ζωή είμαστε αντίπαλοι και σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή στο Μαυροβούνιο. Θεωρώ όμως ότι ο πολιτικός θεσμός αυτός είναι πάρα πολύ ισχυρός στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο, στο πολιτικό κράτος, όχι σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό κράτος. Να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα. Καλούν το ΝΑΤΟ Τρίτο Ράιχ. Υπό κανονικέ συνθήκες, χωρί ε, καμία τιμωρία, χωρίς καμία τιμωρία. Πριν από 15 ημέρες, ε, όχι τότε που γίνονταν οι βομβαρδισμοί, τώρα επιτίθενται κατά των σεξουαλικών μειονοτήτων. Κατευθείαν, άμεσα, δημόσια και συνεχώ. δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το νόμο του Μαυροβουνίου. Δεν ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Είναι εκτό. Ε, κινούνται στα περιθώρια του νόμου. Υφίστανται εκτός του νομικού πλαισίου. Δεν θέλουν να γνωρίσουν το κράτος και να καταχωριστούν. Η Καθολική Εκκλησία έχει καταχωριστεί. Οι Ισλαμικές ε, οργανώσεις είναι καταχωρισμένες. Οι μαυροβουνιακές ε, οργανώσεις έχουν καταχωριστεί. Μόνο η Σερβική Εκκλησία μένει εκτός του πλαισίου του νόμου. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση των σεξουαλικών μειονοτήτων και άλλοι σημαντικοί τομεί στο Μαυροβουνίο. Τι να σας πω, ίσως η Σερβική Εκκλησία τελικά αντιτιθέμενη στις μεγάλες μας αξίες μας προκαλεί να τις προστατεύσουμε και να τις τονίσουμε, αλλά ελπίζω ο πρόεδρος Ντάτσιτς να προάγει τις ε, σχέσεις με, τους, ε, με τις γειτονικέ χώρες, όπου βασικά οι σχέσεις με το Κωσυφοπέδιο είναι βασικό ζήτημα. Συναντήθηκα μαζί τους επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. Τώρα όμως, όπως είπα και σε προηγούμενες δηλώσεις μας, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τη Σλοβανία είναι ότι έχουμε για την Κροατία πλέον πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της Κροατίας και με την υποστήριξη γιατί η Κροατία, ξέρετε, συνδέεται με όλα αυτά τα ζητήματα που ε, πλήττουν τα, Βαλτά, τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι από κοινού θα πετύχουμε μεγαλύτερη ενσωμάτωση και θα μπορέσουμε να καταδείξουμε ότι μπορούμε να καταστούμε ισότιμο μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι μας, και με το Μαυροβούνιο συμπεριλαμβανομένου. President, Αγαπητέ Ράνκο, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση, τη συζήτηση. Η κυρία Λούνατσεκ θα έχει το λόγο αμέσως. Και η συνέχεια αυτής της συζήτησης θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα να, για να μπούμε στις λεπτομέρειες της ενταξιακής διαδικασίας. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ήθελα να υπενθυμίσω στον ε, πρόεδρο ότι δεν μου απάντησε ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στο Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε την κατάσταση για ενδεχόμενη συμμετοχή ενός ποσοστού έως και 30% των γυναικών. Βεβαίως, περισσότερη δημοκρατία στο Μαυροβούνιο και περισσότερες γυναίκες ε, στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο. Το γνωρίζω, το γνωρίζω, έχω πλήρη επίγνωση. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Σας ε, εύχομαι κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο έργο σας.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 meine Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πιέρ Βεμού, εκτελεστικό γενικό γραμματέα της Εξωτερικής Υπηρεσίας, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μας ζήτησε συγγνώμη που καθυστέρησε. Ε, εγώ πρέπει να πω ότι του είπα, του απάντησα ότι κατάφερα να καταφτάσει πολύ, με πολύ μικρότερη καθυστέρηση από ότι η αποστολή στο Μάλι. Είμαστε ευγνώμονες που ήρθε εδώ σήμερα μετά την υπουργική συνάντηση για την ε, υποστήριξη της ομάδας παρακολούθησης και υποστήριξης ε, για το Μάλι σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Μάλι. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε ε, τα πορίσματα της Υπουργική συνάντησης ε, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 5 Φεβρουαρίου με κοινή προεδρία της ΕΚΟΒΑΣ της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΗΕ. Και εμείς είμαστε κάπως ε, απογοητευμένοι γιατί επικρατεί η αίσθηση ότι η στρατηγική που καταστρώθηκε πριν από 2,5 χρόνια για το Σαχέλ δεν έχει πετύχει ιδιαίτερα αποτελέσματα και αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και μετά η αναθεώρηση από πλευρά της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Να μας πείτε ποιες είναι οι αιτίες, γιατί τώρα με το ξέσπασμα του πολέμου τον Ιανουάριο διαπιστώσαμε ότι η απόφαση του Οκτωβρίου να αποσταλούν τα στρατεύματα στο Μάλι δεν ήταν καν σε φάση προετοιμασίας. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια για το τι φταίει. Γιατί όλοι έχουμε συμφέρον τέτοια ζητήματα στο μέλλον να ρυθμίζονται πιο γρήγορα. Και ίσω θα υπήρχε κάποιο τομέα στον οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σα ήμουν λοιπόν ευγνώμων αν θα μπορούσατε στις 31 Ιανουαρίου στο, στη διάσκεψη στη Δόχα συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έγιναν δεσμεύσεις για εκατομμύρια ευρώ. Χαίρομαι που είσαστε εδώ για να μας ενημερώσετε λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ε, thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο λακωνικός, όσο πιο λακωνικός γίνεται. Ίσως συντομότερος και από την αποστολή που έπρεπε να κρατήσει 15 μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω. Θα σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις στο Μαλί. Και θα σας ενημερώσω για τις τρεις διαστάσεις της κρίσης τη στρατιωτική, την πολιτική, διπλωματική και το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης του Μαλή. Θα προσπαθήσω έτσι να απαντήσω και σε μερικές απορίες σας που παρουσιάσετε στα εισαγωγικά σας σχόλια. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική διάσταση, θα ήθελα να πω ότι περνάμε από μία φάση σε άλλη. Τα στρατεύματα του Μαλή και τα στρατεύματα της Γαλλίας έχουν ανακτήσει τις περισσότερες πόλεις του Βορρά με τη βοήθεια των Αφρικανικών δυνάμεων που α, επίσης βοήθησαν. Έχουμε αυτή τη στιγμή επιτόπου 4.000 Γάλλους στρατιώτες ενώ ο στρατός του Μαλή είναι 4 με 5.000 στρατιώτες Έχουμε και αφρικανικές δυνάμεις, 2.000 περίπου στρατιώτες από το Τσάντ και αυτή τη στιγμή αργά αλλά σταθερά φτάνουν και 2.500 στρατιώτες που μετακινούνται προς το βορρά και αναμένονται να γίνουν 5 με 6.000 αργότερα οι δυνάμεις αυτές. Οπότε προχωρεί η στρατιωτική διάσταση. Τώρα όμως αντιμετωπίζουμε μια τελείως καινούργια κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα περάσουμε στη φάση της σταθεροποίησης. Την αποκατάσταση ασφάλειας, όπως λέμε στη στρατιωτική διάλεκτο, την αποκατάσταση ασφάλειας σε όλη τη χώρα και κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου κάποιοι αντάρτες έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή και είναι έτοιμοι να περάσουν την αντεπίθεση με σύντομες τρομοκρατικές επιθέσεις και τέτοιου είδους ε, επιχειρήσεις δημιουργώντας, όπως λέμε στη στρατιωτική διάλεκτο, ένα ασύμετρο πόλεμο, ε, κάτι που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες επί τόπου. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε όλα αυτά. Καταρχήν υποστηρίζει και επιμελητιακά και οικονομικά τις αφρικανικές δυνάμεις, 50 εκατομμύρια από τη διευκόλυνση για την αφρικανική ειρήνη που ανακοινώθηκε στην Αντισαμπέμπα πριν από λίγες μέρες και έχουμε ε, ξεκινήσει την ανάπτυξη της αποστολής EUTN της ευρωπαϊκής δηλαδή αποστολής ε, που θα παράσχει συμβουλές και εκπαίδευση στις δυνάμεις του Μαλή. Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες αποστολές του e UTN Θα συνεχιστεί η άφηξή τους στις επόμενες μέρες. Ε, γύρω στους 500 ε, εκπαιδευτές αναμένεται να αναπτύξουμε και προσωπικό που θα επιληθεί των πρακτικών ζητημάτων και της προστασίας. Μέχρι στιγμής έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και από τις 27 χώρες που έχουν συμβάλει στην επιχείρηση. Η τελευταία χώρα ήταν το Βέλγιο που είπε ότι θα παραμείνουν τα δύο ελικόπτερά του στην περιοχή και θα περάσουν από την γαλλική επιχείρηση στην επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι το κατά πόσο θα προβούμε στην αργή μετάβαση της Αφρικανικής ε, δύναμης υπό την Προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης και της ΕΚΟΒΑΣ και τη μετατροπή της σε μια αποστολή αποκατάσταση της ειρήνης ε, των Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά για τη μετάβαση αυτή χρειάζεται κάποιος χρόνος και χρειάζεται και συμφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να εγκριθεί ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα καθορίζει την εντολή και το έβρος της αποστολής αυτής ε, της ειρηνευτικής δύναμης και επίσης και τις πρακτικές λεπτομέρειες αυτής της ειρηνευτικής δύναμης. Και επίσης ποια θα είναι η εξέλιξη. Παρόλο που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της δύναμης του ΙΕ θα περιλαμβάνει ε, της, ε, ένα μεγάλο τμήμα των αφρικανικών δυνάμεων. Τώρα, για τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσεις ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σταθερότητας ε, στο στρατιωτικό τομέα ώστε να μπορέσει η ειρηνευτική δύναμη να αναλάβει. Όπως είπε ο Μπάνκι Μουν, για να υπάρξει μια αποστολή αποκατάστασης ειρήνης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ειρήνη κάτι που δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη αξιολόγηση κατάστασης που θα πρέπει να γίνει πριν περάσουμε στη μετάβαση σε μια ε, ειρηνευτική δύναμη, σε μια δύναμη ε, διαφύλαξης ε, της ειρήνης. Οπότε μια τέτοια διαδικασία θα είναι μελλοντική. Προς το παρόν εξακολουθούν να ισχύουν οι άλλες ρυθμίσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μπαμάκο, και αυτό είναι το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, αυτή τη στιγμή στον Μπαμάκο η πολιτική κατάσταση είναι αρκετά ήρεμη και ο πολιτικός οδικός χάρτης έχει εγκριθεί με δύο πτυχές, με δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την πολιτική διαδικασία που θα καταλήξει στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου και μάλιστα η ημερομηνία για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών θα είναι η 7η Ιουλίου, μόλις έχει ανακοινωθεί. Μερικοί παρατηρητές θεωρούν ότι παρά είναι φιλόδοξη αυτή η ημερομηνία. Πάντως τουλάχιστον έχει καθοριστεί. Ε, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις αρχές του Μαλή ώστε να τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, ε, έναρξη μιας διαδικασίας επανασυμφιλίωσης και εθνικού διαλόγου με τη σύσταση μιας Εθνικής Επιτροπής που θα εξετάσει και θα προσπαθήσει να φέρει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλες τις κοινότητες και από το Βορρά και από το Νότο και όχι μόνο τις κοινότητες του ΑΡΕΓ αλλά και τους υπόλοιπους. Αυτή η διαδικασία ίσως προσκρούσε σε δυσκολίες γιατί δεν έχει οριμάσει ακόμη η κατάσταση. Πάντως κάποια στιγμή η διαδικασία αυτή θα συνδυαστεί και με την ε, εκλογική διαδικασία γιατί θα πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μερικοί στον Παμάκο λένε ότι καμία λύση επανασυμφιλίωσης δεν πρόκειται να βρεθεί αν δεν αναλάβει νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ώστε να δώσει να μιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία επανασυμφιλίωσης. Και εμείς ε, υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία με οικονομική αρρωγή αλλά και τεχνική αρρωγή που θα χορηγήσουμε στις ε, αρχές του Μαλή και επίσης θα δώσουμε τεχνική υποστήριξη και για την εκλογική διαδικασία και φυσικά θα στείλουμε αποστολή παρατήρησης εκλογών εν το χρόνο δεν έχουμε χάσει χρόνο ως προς τα θέματα της οικονομικής ε, συνδρομής. Βοηθούμε το Μαλί με βραχυπρόθεσμη οικονομική αρρωγή μέσω του μέσου σταθερότητας 20 εκατομμύρια ε, βοήθεια στο πακέτο προκειμένου να βοηθήσουμε τις απελευθερωμένες ζώνες του Βορρά να αποκαταστήσουν ε, τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, που επιλήγησαν τον τελευταίο καιρό, να βοηθήσουμε στην εκλογική διαδικασία και σε ορισμένα άλλα θέματα. Όπως ανήγγειλε ο Επίτροπος Πίμπαλξ, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα αρρωγής ε, που είχε παγώσει για ένα διάστημα για ένα πακέτο 250 εκατομμύριων ευρώ προκειμένου να βοηθήσουμε το Μαλί ε, να υλοποιήσει τις προτεραιότητες ε, επιστηστικής ασφάλειας, υγείας, ε, εκπαίδευσης και μάλιστα το συντομότερο δυνατό να περάσουμε και σε μία δημοσιονομική υποστήριξη ώστε να βοηθήσουμε την ανοικοδόμηση του κράτους του Μαλή το συντομότερο δυνατό. Να προσθέσουμε και την ανθρωπιστική ενίσχυση πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια και το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Εκεί έχουμε μια, με όλα αυτά έχουμε μια καλή εικόνα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί. Βέβαια, μερικοί θα πούν ότι α, είναι κάπως καθυστερημένα όλα αυτά, αλλά σας διαβεβαιώ ότι οι αρχές του Μαλί δεν συμφωνούν με αυτή την επίκριση. Ο Πρωθυπουργός του Μαλί έχει δηλώσει επανειλημμένω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο βασικό υποστηρικτή και ο κύριο εταίρο σε όλη τη διάρκεια τη κρίση από την αρχή. Και μάλιστα μερικέ φορέ ξεχνούμε ότι μία από τι δυσκολίε που αντιμετωπίσαμε στην ε, σύσταση και την ανάπτυξη της EUTN ήταν ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε ένα πραξικόπημα στο Μαλί που οδήγησε στην κατοχή της μισής επικράτειας της χώρας και χρειάστηκε αρκετό διάστημα για να μπορέσουν οι συνταγματικές αρχές, οι νόμιμες αρχές της Μπαμάκο να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και να μας δώσουν το πράσινο φως για να περάσουμε στην εφαρμογή της e UTN της Ευρωπαϊκής Αποστολής. Και μόνο τον Ιούλιο-Αύγουστο προσωρινός πρωθυπουργός επέστρεψε στο Μαλί, σύστησε την κυβέρνηση και έκτοτε εμείς ε, προχωρήσαμε με ταχύς ρυθμούς για την ανάπτυξη της EUTN και μάλιστα επιταχύναμε την διαδικασία ανάπτυξης ε, ε, της EUTN από το ξέσπασμα της κρίσης τον Ιανουάριο και καταφέραμε τα τα πρώτα τμήματα της UTN να τα αναπτύξουμε μέσα σε ένα μήνα. Θα μπορούσαν να πούν κάποιοι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο γρήγοροι, αλλά σας διαβεβαιώ ότι επί τόπου όλοι είναι ευτυχείς που έχει αναπτυχθεί η UTN και άρχισε να εργάζεται το συντομότερο δυνατόν. Λυπούμε λοιπόν, αν μακρηγόρησα, θα σταματήσω λοιπόν εδώ προς το παρόν. Thank you very much, Pierre, for... Σας ευχαριστούμε, Πιέρ, για την πληροφορίες αυτές, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λάκη. Ευχαριστώ κύριε Δημόντ, μας δώσατε μια εικόνα μιας περίπλοκης κατάστασης. Είναι εντυπωσιακή η κατάσταση από πλευράς ανθρωπιστικής, οικονομικής επιμελητίας, αλλά και σε ό,τι φάει μακροπρόθεσμη βοήθεια. Μιλάμε για ένα πακέτο περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Αν ε, βάλουμε τα 250 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική μακροπρόθεσμη βοήθεια, 20 εκατομμύρια πακέτο στήριξης για τον ε, Βορρά και 50 εκατομμύρια για θέματα επιμελητίας. Ε, εντυπωσιακό ποσό για, το, για την έκταση της, του Μαλή και για την έκταση της κρίσης. Αυτό που μας λείπει είναι η πολιτική εικόνα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Αλγερία, το ρόλο της Αλγερίας. Αν πραγματικά δεν θέλουμε να στρουθοκαμιλίζουμε και να λέμε ότι η λύση του στο Μαλί έχει επιληθεί με την γαλλική παρέμβαση και αν κατανοήσουμε την εικόνα στο Σαχέλ χωρίς ε, την εμπλοκή της Αλγερίας και χωρίς πλήρη αλλαγή των πολιτικών, της πολιτικής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέμα, θέματα ε, συγκαλυμμένων ενεργειών και μυστικών υπηρεσιών και όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε πολλά. Όπως ξέρετε, οι τρεις βασικές ομάδες εκεί, οι μαφιόζικες, ε, τρομοκρατικές οργανώσεις όπως τις ε, αποκαλώ, γιατί έχουμε πρώτης ε, τάξης ε, μαφιόζικες οργανώσεις και τρομοκρατικές οργανώσεις, υποστηρίζονται τα τελευταία χρόνια μυστικά, ίσως και όχι τόσο μυστικά από την Αλγερία, με την ε, συνένεση των δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Και οι ομάδες αυτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όπως έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο και έχουν χρηματοδότηση και όταν καταλαβαίνει, όταν καταλαβαίνει όταν καταλάβουν πια ότι δεν έχουν την υποστήριξη την οποία είχαν στο παρελθόν. Άρα, χρειαζόμαστε σαφείς ιδέες για το τι θα πρέπει να γίνει στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Αλγερία. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να σημειώσουμε μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ και θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον ε, κύριο Βημών. Εγώ είμαι από τους μεγαλύτερους ε, θαυμαστές σας. Οι τζιχάντι, οι τρομοκράτες αποτελούν απειλή για την περιφέρεια και πέραν αυτής. Ε, και αν δεν τα καταφέρει το Μαλί, τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος, αποτέλεσε ε, άμεση δικαιολογία για να παρέμβει ο πρόεδρος Ολάντ και οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Και η οξία φάση του πολέμου έφτασε σε μία, οδήγησε σε μία νίκη, αλλά υπάρχει μία τάση ασυμμετρίας και επαναφοράς ε, ε, τουλάχιστον ασύμετρων στρατιωτικών σειράξεων και στο Μπαμάκο και στο Νότο οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις θεωρούνται ως ελευθερωτές. Αλλά αυτοί που συνεργάστηκαν με τη Τζιχάντ και άλλες δυνάμεις, δεν θυμάμαι και το άλλο ακρόνιμο, όλοι αυτοί ίσως έχουν μεγάλες, μεγάλα αντίπεινα από τοπικούς παράγοντες που εφαρμόζουν τη Σαρία. Εμείς υποστηρίζουμε την ταχεία επέμβαση της Γαλλίας και καλωσορίσαμε και τη συμμετοχή της δικής μας χώρας και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μία διμερής ή τριμερής, ένα διμερές ή εγχείρημα και φαίνεται όταν μιλάμε για ταχεία επέμβαση ότι μπορεί να γίνει από δύο χώρες κυρίως, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν ε, συμμετέχουν το ΝΑΤΟ ή άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ως προς την κατάσταση τώρα και την τρομοκρατική απειλή Πού πιστεύετε, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση και ο, ο έχει κοιτάσματα ε, ουρανίου και οι τρομοκράτες μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα ορυχεία. Θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα στόχο τον οποίο θα πρέπει να υπερασπιστούμε. Οι στρατιωτικοί κύκλοι μας είπαν ότι δεν έχουν εντολή να προστατεύσουν τον Ήγυρα ή τα κοιτάσματα ουρανίου, τα ορυχεία ουρανίου. Νομίζετε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε, να οδηγήσουμε στην οικοδόμηση αυτών των χωρών τη στιγμή που υπάρχουν σύνορα τα οποία είναι εύκολα διαβατά. Μπορεί να, ε, γίνουν, να μεταφερθούν ναρκωτικά όπλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Θεωρείτε τώρα ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μία ε, ζώνη ασφαλείας στην περιοχή του Σαχέλ, γιατί εγώ συντάσω μία έκθεση Έχουμε έξι ομιλητές. Προσπαθήστε να ε, επιταχύνετε. Ε, Γκάλερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση για την ε, αποστολή εκπαίδευσης. Στη Σομαλία έχουμε κάποιες σχετικές ε, εμπειρίες σε ό,τι αφορά την αλυσίδα πληρωμής η οποία δεν τηρήθηκε και τελικά οι εκπαιδευόμενοι στράφηκαν αλλού. Έχουν διευκρινιστεί αυτά με τις αρχές του Μαλή και είναι σε θέση οι αρχές του Μαλή να πληρώσουν τους στρατιώτες. Ούτε να λαμβάνουμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και επίσης το ερώτημα το εξής. Ποιον εκπαιδεύουμε συγκεκριμένα. Ένα τμήμα του στρατού ε, έκανε το πραξικόπημα. Αποτελούν και αυτοί ε, άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν την εκπαίδευση. Είναι οι άλλοι, είναι όλοι μαζί. Είναι αυτό το τμήμα της εθνικής συμφιλίωσης ε, στο ιστορικό του στρατού. Και πώς εξασφαλίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα τηρηθούν στο πλαίσιο αυτό. Γιατί ακούσαμε ότι ο στρατός έχει κάνει επιθέσεις ε, στους Τουαρέγ. Ευχαριστώ. Κυρία Νάτς. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέ. Σας ε, ευχαριστώ θερμά που ήρθατε για να μας ε, παρουσιάσετε αυτή την περιστατωμένη εικόνα της κατάστασης γιατί εδώ και τέσσερις εβδομάδες ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση αν μετράω σωστά και ήδη μας δώσετε μία πλήρη επισκόπηση της κατάστασης που είναι καθησυχαστική από κάποια άποψη και από άλλη όχι τόσο. Και οι λιγότερο εφησυχαστικές πτυχές αφορούν το κίνδυνο μετατροπής της σύγκρουσης αυτής από μια κλασική στρατιωτική σύγκρουση, κάτι που είχε μέχρι τώρα, σε μια σύμμετρη σύγκρουση. Ε, κάτι που θα ε, δημιουργήσει την πιο ύπουλη και ολέθρια μορφή εχθροπραξιών με θύμα το, το λαό. Απευχόμαστε οπωσδήποτε μια τέτοια εξέλιξη και μετατροπή αυτής ε, της σύγκρουσης. Ο κύριος Αρλάκη είναι πολύ πιο δεξιοτέχνης και πολύ πιο τώρα από μένα Α, πιστεύω παρόλα αυτά ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε, να διατηρήσουμε να αναπτύξουμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και τους κοντινούς γείτονες, την Αλγερία δηλαδή, το Μαρόκο, τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη, την Ιγυρία, τον Ήγυρα και με τους ε, πιο απόμακρους γείτονες. Έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες με, ποιους, με ποιο τρόπο. Πρόσφατα στο Ραμπάτ μάθαμε με κάποιους συναδέλφους ότι η ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την κατάσταση ασφάλειας ε, αποκαταστάθηκε τελικά μεταξύ της Αλγερίας ε, και του Μαρόκου, αλλά πολύ πρόσφατα. Άρα θα πρέπει να ενταθούν εκεί οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ανάμιση και αυτών των χωρών. Μπορείτε να μας δώσετε λίγες πληροφορίες για το τι συμβαίνει εκεί. No, it's now Mr. Bicep. Oui, merci. Euh, ce que je voulais... Θα ήθελα να πω, με βάση αυτά που είπατε, μιλήσατε για εθνική συμφιλίωση, η οποία είναι απολύτως αναγκαία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εξευρεθούν εταίροι για διαπραγμάτευση. Και για να βρεθούν εταίροι θα πρέπει να δεχτούμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων εκείνους ε, οι οποίοι συμμετέχουν στις σειράξεις. Μιλώ για το MLNA. Ξέρετε ότι στο Βόρα υπάρχει ε, ένα πόσμασμα του MLNA το οποίο δρά επιτοπίως, το αναφέρει και ο τύπος και γίνεται λόγος για αυτό το κίνημα. Και ξέρω ότι υπήρξαν εντάλματα σύλληψης κατά μελών του ΕΜΕΛΕΝΑ. Εάν θέλουμε λοιπόν να βρούμε τέρους θα πρέπει καταρχήν να μην υπάρχει ποινικοποίηση. Δεν θα βρεθεί και ούτε καν στρατιωτική λύση. Μας μιλήσατε και για ένα χρηματοοικονομικό σκέλος για την ανασυγκρότηση και ασφάλεια αυτής της χώρας. Αλλά όποια χρηματοδοτική προσπάθεια και να κάνουμε για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας, εάν δεν προϋπάρξει πολιτική συμφωνία, τότε όλα θα είναι σαφρά θα πρέπει να φτάσουμε σε μια πολιτική συμφωνία με βάση την κατάσταση των συνόρων όπως αναγνωρίζονται διεθνώς και θα πρέπει και οι γείτονε χώρες να συμμετέχουν σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Ο κύριος Ευχαριστώ και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και για τις πληροφορίες. Η ομάδα μου στην Ολομέλεια ε, καταφέρθηκε κατά της, παρέμβασης, της επέμβασης της Γαλλίας γιατί θεωρούμε ότι οι, οι δεν είναι ούτε Βέρβεροι ούτε Άραβες και γι' αυτό θα πρέπει να τους υπερασπιστούμε μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ανεξαρτησίας και από τότε που δρούσαν οι απικιοκράτες στην περιοχή είχαν αποκλειστεί και θεωρήθηκαν διαφορετική κατηγορία από τους ε, Βερβέρους. Και άρα η εξέλιξη της στρατιωτικής επέμβασης ήταν ε, ε, περίεργη. Τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Ολάντη είπε ότι δεν θα επέμβει. Τον Ιανουάριο είπε ότι θα επέμβει περιορισμένα ενώ ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας είπε ότι ο στόχος είναι να ανακατακτήσουμε το Μάλι. Και επειδή υπάρχει σύγχυση στόχων, χρησιμοποιήθηκαν ε, πολλά επιχειρήματα, δηλαδή ότι οι σαλαφιστές τι κάνουν, εφαρμόζουν τη σαρία στο Τιμπουκτού και κόβουν χέρια και προβαίνουν σε ακραίες ποινές. Και με τη βοήθεια του Κατάρ δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ στην ε, περιοχή του Σαχέλ. Είναι οι ίδιοι τους οποίους όπλησε το Κατάρ κατά του δικτάτορα Καντάφη. Αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται επίσης και στη ε, περιοχή του Ασαουάντ. Αυτή η αμφισημία είναι αντιφατική. Και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία του σαλαφισμού θα μας ε, οδηγήσει σε ένα δρόμο χωρίς ε, ε, διέξοδο. Και εν πάση περιπτώσει η παρέμβαση του Κατάρ είναι κάτι το αρνητικό. Στην στρατιωτική επέμβαση, κατά τη στρατιωτική επέμβαση δεν γίνεται λόγος για την όμορφη περιοχή με το ε, Νίγηρα, διότι η Γαλλία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά κοιτάσματα ουρανίου που ενδιαφέρουν τη Γαλλία και είναι περιοχή που θέλει να ελέγξει η Γαλλία ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα ουρανίου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Ο κύριος Αρλάκη μίλησε για την Αλγερία και θα προσπαθήσω να απαντήσω και στο ερώτημα που, εθίγει για, την για όλη την περιοχή τι θα κάνουμε. Η Νέτσερ και Τάνοκ αναφέρθηκαν σε αυτό. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα του Μάλι θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα της περιοχής του Σαχέλ και όλες οι όμορες χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν. Εξ ονόματος της ε, είπα της εκπροσώπου, μία εβδομάδα πριν στο Παρίσι παρευρέθηκα σε μία σύνοδο για, που αναφερόταν στη Λιβύη, στην κατάσταση της δικαιοσύνης και από την Τρίπολη μου είπε ο πρόεδρος, ο υπουργό με συγχωρείτε εξωτερικών, ότι δεν θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα εάν δεν δούμε πώς το αντιμετωπίζουν και οι όμορες χώρες, διότι οι επικεφαλής κρατών δεν θα σας μιλήσουν μόνο για το Σαχέλ. Μιλώ για τον Νίγηρα, τη Μαυριτανία, την, ε, το Μαλί μιλούν και για τη Σομαλία, ακόμα και για την Κεντρική Αφρική, διότι η τρομοκρατική δράση αυτή, η δράση της μαφίας, διαχέεται από τη, τη δυτική πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Και ακόμα και αν οι Αλγερινοί δεν ήταν τόσο θετική και μετά την τρομοκρατική, το τρομοκρατικό συμβάν στην Αλγερία, βλέπετε ότι δεν μπορούσαν να ε, αντιδράσουν διαφορετικά βλέπουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα δίκτυο πληροφοριών για τους ε, τρομοκράτες και σε εκείνη την περιοχή προέρχονται από ένα πιο διάχυτο κίνημα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχοληθήκαμε με αυτή τη στρατηγική για ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ και γι' αυτό και η Αφρικανική Ένωση ζήτησε κάτι παράλληλο. Και οι Ρωμάνο Πρόντι και Μπάνκι Μουν αυτό ακριβώς ε, προσπαθούν να προβλέψουν. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τις διαφορές περιφερειακές οργανώσεις, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπλεκόμενες χώρες θα πρέπει να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να συγκρίνουμε τις πληροφορίες μας για να καταπολεμήσουμε, καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Για να φτάσουμε στη ρίζα της κακοδαιμονίας, το λαθρεμπόριο, το εμπόριο ανθρώπων και οποιοδήποτε είδος ε, λαθρεμπορίου ή παράνομης εμπορίας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και πρόκληση συνάμα. Για να απαντήσω στον κύριο Τάνοκ, ακόμα και εάν αυτές οι τρεις βασικές ομάδες ε, που βρίσκονται στο Βόρειο Μαλί έχουν Ακόμα και αν αυτές οι τρεις ομάδες έχουν πληγεί από τις γαλλικές δυνάμεις και ιδιαίτερα εισάλτη περισσότερο από τις δύο άλλες, υπάρχουν, είναι ανθεκτικές ομάδες και θα μπορέσουν να αντεπιτεθούν. Θα πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό και να συνεργαστούμε για να βρούμε το κατάλληλο δρόμο αντιμετώπισης. Αυτό είναι κάτι το μακροχρόνιο, μία μακροχρόνια στρατηγική. Και εσείς κύριε Τάνοκ αναφερθήκατε ε, στον Νίγηρα. Δεν, είναι, δεν πρόκειται το ίδιο για, το, για την ίδια σχέση που υπάρχει με το UTM. Ε, στην περίπτωση του Νίγηρα, του άκρου αυτού, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης των ε, τρομοκρατών. Πρόκειται για την στρατιωτική αποστολή αυτή, την UTM, για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι, δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει και στο Νίγηρα και στο ε, Κέρας και στην Αλγερία γιατί πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία και θα πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Γιατί δεν δράσαμε τόσο γρήγορα όσο η Γάλλοι, μα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ακόμα κι αν ε, είχαμε ε, ετοιμοπόλεμες ε, δυνάμεις, ξέρετε ότι οι ετοιμοπόλεμες μονάδες δεν μπορούν να κινητοποιηθούν σε 24 ώρες, χάρη ένας μήνας, έξι εβδομάδες. Γιατί οι Γάλλοι έδρασαν άμεσα. Γιατί είναι οι μόνοι στη Δυτική Αφρική που έχουν δυνάμεις στη Σενεγάλη, στο Τσάντ και στην, ε, και στην ακτή του Ελεφαντοστού. Μπόρεσαν λοιπόν να βρεθούν εκεί επιτόπου άμεσα. Εμείς όμως ως Ευρώπη δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να το κάνει. Το ζήτημα είναι ποιος έχει την ικανότητα να δράσει άμεσα γιατί ξέρετε ότι μας καταλάβανε εξαπίνης αυτές οι δυνάμεις. Στην Πορκίνα Φάσο είχαμε διαπραγματεύσεις με την MNLA την Κυριακή για μια πολιτική λύση. Έφυγαν από το τραπέζι, ε, αποχώρησαν και άρχισαν με τη στρατιωτική επέμβαση. Αν αυτό δεν θεωρείται έκπληξη δεν ξέρω τι είναι, τι θεωρείται. Χρειαζόταν λοιπόν άμεση επέμβαση, μια άμεση αντίδραση και λίγες χώρες είχαν αυτή τη δυνατότητα. Χρειαζόταν λοιπόν και έγινε η ταχεία επέμβαση από τις γαλλικές δυνάμεις, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε υπομορφή προστιθέμενης αξίας, διότι η στρατιωτική ικανότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διπλωματία, από την ανθρωπιστική βοήθεια και από τα αναπτυξιακά προγράμματα. Περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για συνεκτική δράση. Αυτό ακριβώς κάναμε και στο κέρας της Αφρικής και τη Σομαλία. Κύριε Γκάλερ, για τη Σομαλία είπατε κατά πόσο η UTM θα μπορούσε να αποτρέψει ορισμένες δυσκολίες, όπως ίσχυσε στην περίπτωση της Σομαλίας και της Ουγκάντας. Θα τα καταφέρουμε, γιατί στην περίπτωση του Μάλι δεν ε, μιλάμε για την ίδια κατάσταση όπως επικρατούσε στη Σομαλία που δεν υπήρχε κυβέρνηση, γιατί εδώ δεν υπήρχε κυβέρνηση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μεταβατικός πρόεδρος είναι ο πρώην επικεφαλής της ε, Εθνικής Βουλής. Γι' αυτό θα πρέπει να αναμείνουμε τις εκλογές. Πρόκειται για μία νόμιμη αρχή έναν πρόεδρο που ζήτησε τη διεθνή βοήθεια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυβερνά τη χώρα, υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών και άρα δεν είναι δύσκολο να προχωρήσει και το χρηματοδοτικό σκέλος, να διοχετευτεί προς τα εκεί. Συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για αναδιάρθρωση του στρατού του Μάλι, έτσι ώστε να είναι πραγματικά ε, ένας εθνικός στρατός. Αυτό είναι μία μακρόπνοη διαδικασία, αλλά α, ακριβώς αυτό θέλει να κάνει ο στρατηγός Λεκουάντρ. Εκπαιδεύει τις ένοπλες δυνάμεις Πρόκειται για μία διαδικασία εκπεριτροπής, αλλά συμβουλεύει και το στρατό για την επαναδιοργάνωσή του, πώς μπορούν να ενταχθούν οι, διάφορες εθνοτικές κοινότητες, έτσι ώστε να έχουμε έναν εθνικό στρατό που να είναι πραγματικά εθνικής εμβέλειας. Η κατάρτιση των ενόπλων δυνάμεων έχει μεγάλη σημασία και με στα πλαίσια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, των ΜΚΟ και των παρατηρητών από την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, που επιτοπίως θα δουν τι συμβαίνει στις διάφορες πόλεις ως προς την παραβίαση, ενδεχόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Μπισέπ, μιλήσατε για την ε, εθνική συμφιλίωση. Ας μιλήσω και γαλλικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί έγκυται η πεμπτουσία του προβλήματος. Και υπάρχει πρόβλημα με το MNLA, διότι το MNLA για μεγάλο χρονικό διάστημα μίλησε για μία ανεξαρτησία του Σαουάντ, δηλαδή της περιοχής που ζουν οι Τουαρέγ και αμφισβητεί την, ε, την ε, επικράτεια, την εδαφική ακαιρεότητα του Μάλι. Οι αρχές του Μάλι λοιπόν δεν μπορούσαν παρά να μιλήσουν με ομάδες και κοινότητες που δέχονται αυτή την εδαφική ακαιρεότητα και το σύνταγμα του Μάλι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και η αντιπροσωπεία μας ε, επιτόπου προσπαθεί ακριβώς αυτό να κάνει. Ε, είναι μία μακροχρόνια διαδικασία και αυτή η διαδικασία εθνικής ε, επανασυμφιλίωσης δεν είναι εύκολη. Μιλήσατε για συλλήψεις. Ναι, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό εκ του σύνεγγης. Μας ενδιαφέρει μία διαδικασία νομιμότητας και δικαιοσύνης και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόκειται για μια διαδικασία που θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί αυτή τη στιγμή κατέχουν το Κιντάλ οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν σε ένα κοινό εγχείρημα με το Τσάντ υπάρχουν κοινέ δυνάμεις και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό με τις αρχές του Μπαμακο. Μπαμάκο. Κύριε Μέιρ, μας είπατε ότι η φυλή των Τουαρέγκ είναι μια παλαιά μακραίωνη φυλή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά η λύση δεν μπορεί να είναι στρατιωτικής υφής, μόνο πολιτικής. Αυτό ακριβώς προανέφερα. Δεν είναι εύκολο, χρειάζεται χρόνος, αλλά αν δείτε τι έγινε στον Νίγηρα και πώς προοδευτικά επέλυσαν το θέμα των Τουαρέγ, ε, αυτό ακριβώς μας καταδεικνύει ότι υπάρχει πείρα σε αυτό το τομέα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. κυρία Γκόμες για το λόγο καταρχάς και άλλοι δύο συνάδελφοι. Η κυρία Γκόμες λοιπόν, Λουράτα και Λουζέν. Κυρία Γκόμες, έχετε λόγο. Θα ήθελα κύριε Δημότ να σας ρωτήσω το εξής. Στο τελευταίο Συμβούλιο συζητήθηκαν θέματα χρηματοδότησης για την αποστολή ΚΕΠΑ, όπως ε, η αποστολή στο Μαλί. Δεν ε, αποτελεί αυτό ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αποστολές αυτές. Ένα θέμα είναι η έλλειψη συγχρηματοδότησης. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν την ευκαιρία αυτή. Όχι μόνο λόγω της γαλλικής ε, πρωτοβουλίας, αλλά και λόγω της ε, απειλής για την δική μας ασφάλεια σε ό,τι αφορά το τμήμα αυτό, αλλά και άλλα τμήματα της Αφρικής. Να ρωτήσω επίσης το εξής. Πείτε μας, αν θέλετε, ποια είναι η σχέση που έχουμε με την ΕΚΟΒΑΣ και την Αφρικανική Ένωση. Έχουμε δώσει τόσα πολλά χρήματα ε, στο μέσο αυτό για την ειρήνευση στην Αφρική. Θεωρείτε ότι υπάρχει αποτέλεσμα για τον πολιτικό τώρα συντονισμό στο Μαλί και στην όλη περιφέρεια. Ξέρουμε ότι τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται στο κέρας της Αφρικής όταν ε, πετύχαμε ακριβώς τον πολιτικό συντονισμό αυτό. Έχουμε υπόψη κάποιο τέτοιο πολιτικό συντονισμό με την UTM ε, για το Μαλί, για την πολιτική ε, ειρήνευση, για την εκλογική διαδικασία, για την οικοδόμηση θεσμών και για την ευρύτερη περιοχή. Αναφερθήκατε στη Λιβερία, στον Ήγηρα κτλ. Τέλος. Ό,τι και να πιστεύουμε ότι αποτελεί ότι είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις που πολεμάμε. Ξέρουμε που χρηματοδοτούνται. Τα παίρνουμε λοιπόν σοβαρά τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για οικονομικά θέματα, αλλά για ανθρωπιστικά. Μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4.000 Γάλλους στρατιώτες. Ξέρουμε ότι ο Γαλλικός στρατός δεν θα παραμείνει στο Μαλί, αντίθετα με ό,τι ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Και ξέρουμε ότι έχουμε 5-6.000 στρατιώτες ε, από το Τσάτ και την Αφρική. Μας είπατε επίσης ότι 500 είναι το προσωπικό της EUTN, εκ των οποίων 200 είναι εκπαιδευτές. Πώς θα διασφαλίσουμε λοιπόν την ασφάλεια στο Μαλί εφόσον θα, φύ, θα εγκαταλείψει το Μαλίο Γαλλικό στρατός ε, και πρώτα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους Αφρικανούς στρατιώτες. Τι θα γίνει με την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίφαση ασφάλεια στο Μαλί χάρη στην παρουσία των ε, γαλλικών στρατευμάτων. Από τη στιγμή που θα ε, αποχωρήσουν, πώς θα γίνει ο συντονισμός μεταξύ της εκπαίδευσης και της ανάληψης της αποστολής. Θα προλάβετε εγκαίρως να εκπαιδεύσετε τους Αφρικανούς στρατιώτες. Ευχαριστώ κυρία Λέζινγκ. Θα ήθελα να κοιτάξουμε και πάλι τις διαπραγματευτικές δυνατότητε για το μέλλον. Να κάνω κάποια ερωτήματα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάντα πολύ επικίνδυνο σε μια κατάσταση στρατιωτικής ε, επέμβασης, παρέμβασης, παρά το γεγονός ότι εκφράστηκε διαφορετικά αυτό. Η διπλωματική παρέμβαση και η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ουσιαστικά υπονομεύονται. Και όταν κοιτάμε παλαιές συγκρούσεις στη Λιβύη, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι εκεί ένα πρόβλημα ήταν ότι έγινε στρατιωτική παρέμβαση χωρίς να υπάρχει ένα όραμα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι Υπήρξε και σχετική εμπλοκή και των ε, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην Αλγερία, τις οποίες τις χειρίζεται ο Λίβανος. Γι' αυτό λοιπόν, η Λιβρία, θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη αυτά. Συγκεκριμένα, ρωτώ το εξή. Συμφωνούμε ότι μιλάμε για μια σύγκρουση που διαρκεί επί δεκαετίες. Το αναφέρετε κι εσείς αυτό. Δεν άκουσα όμως να μας πείτε ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης υπάρχουν. Για παράδειγμα, στη δεκαετία των 90 υπήρξε σχετικός ε, πόλεμος, έγινε ειρηνευτική συνθήκη μετά που προέβλεπε πληρωμές από τον πιο πλούσιο νότο προς το βορρά οι οποίες όμως δεν συνεχίστηκαν οι πληρωμές αυτές από πλευράς του νότου. Τι γίνεται, θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί μία δυνατότητα για το μέλλον δεν μπορούμε να πούμε ότι «Α, κοιτάξτε, πρόκειται για επαναστάτες και δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους γιατί δεν σέβονται το Σύνταγμα». Είναι πολύ διαφορετικοί οι επαναστάτες. Και είναι και επαναστάτες που δεν είναι μόνο Ισλαμιστές. Ένα άλλο ερώτημα σε ό,τι αφορά ανθρωπιστικά και στρατιωτικά θέματα. Είδα μια εκπομπή στην τηλεόραση όπου αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει καμία πρόσβαση για δημοσιογράφους στην, στην εμπόλεμη ζώνη. Αυτό είναι προβληματικό και για τη δημοκρατία, αλλά και οι δημοσιογράφοι δήλωσαν ότι και για αυτούς δεν ε, ήταν δυνατόν να μεταφούν στις περιοχές αυτές. Φοβούνταν για τη ζωή τους, γιατί οι αεροπορικές επιθέσεις θα είχαν θύματα χωρίς διακρίσεις. Ποιος είναι λοιπόν ο εχθρός όταν κάνουμε πολεμικές, ε, πολεμ, ε, αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αν κινδυνεύουν δημοσιογράφοι, θα κινδυνεύουν και άλλα άτομα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τους ε, Ισλαμιστές, με τη μαφία, με την τρομοκρατία. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα ενισχυμένης αυτονομίας σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση της περιοχής των Τουαρέγ ή το θέμα είναι να επανέλθει η κατάσταση στο πώς ήταν προηγουμένως. Κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, μπορούμε να κάνουμε πόλεμο με δίκαιο τρόπο για τους δημοσιογράφους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος γιατί ο χρόνος πιέζει. Κυρία Γκόμες, θα σας απαντήσω στα γαλλικά, μια και θέσετε την ερώτηση στα γαλλικά. Oui, Για τη χρηματοδότηση. Ναι, θα γίνει όπως και το υπόλοιπο με βάση εθνικές συνεισφορές. Δεν είναι άλλωστε από τις πιο ακριβές επιχειρήσεις, από τις πιο δαπανηρές επιχειρήσεις που είχαμε στα πλαίσια της α, ε, κοινής πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας και άλλες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο δαπανήρες. Ε, η αφισμά, για παράδειγμα, είναι πιο δαπανήρη. Τώρα, αν θα είναι αποδοτική αυτή η αξιοποίηση των κονδυλίων, μα κοιτάξτε, αν δούμε που βρίσκεται η Σομαλία σήμερα, μετά από δέκα, χρόνια και ό,τι προσπάθεια έγινε, έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρόοδος έγινε, έγινε χάρη σε εμά και για την καταπολέμηση της πειρατείας και για την υποστήριξη της αφρικανικής δύναμης και για την ε, εκπαίδευση των ε, δυνάμεων της ε, ελίτ, δυνάμεων ελίτ της Αφρικανικής Ένωσης. Νομίζω ότι πραγματικά τα χρήματα στη Σομαλία αξιοποιήθηκαν πλήρως, ε, δεδομένη της πρόοδου που σημειώθηκε και της, ε, του φόρου τιμής που αποτείουν, από, που αποτείουν όλοι στην Ευρώπη που πραγματικά πρωτοστάτησε στις επιχειρήσεις στη Σομαλία. Εκτός μικροφόνο δυστυχώς ε, το σχόλιο της κυρίας Γκόμες. Με το African Peace Facility ε, χρηματοδότησε κυρίως την Αμισόν και ε, θα χρηματοδοτήσει τώρα την Αφίσμα, την νέα αφρικανική δύναμη που θα αναλάβει στο Μαλί. Και νομίζω ότι είναι μια καλή χρήση των κονδυλίων μας καλύτερα να τα τοποθετήσουμε τα κονδύλια αυτά στην αφήσμα στην Αφρικανική Δύναμη που θα αναλάβει το έργο της σταθεροποίησης στο Μάλι. Επίσης θα διορίσουμε έναν ειδικό εκπρόσωπό μας για το Σαχέλ. Είπατε εκπρόσωπος θα ορίσει κάποιον τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, δεν ξέρω και ελπίζω να είναι εξίσου επιτυχημένη η αποστολή του με αυτή του αντίστοιχου αντιπροσώπου στο κέρα τη Αφρικής. Και θα είναι χρήσιμο για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως να διορίσουμε και τέτοιο ειδικό εκπρόσωπο, γιατί χρειαζόμαστε και μία ένταση προσπάθειας στην περιφερειακή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για, για τα στρατεύματα που παρίστανται στην περιοχή αν αποχωρήσουν τα γαλλικά στρατεύματα όπως ανήγγειλε η Γαλλία θα αφήσουν στο πόδι τους μία αφρικανική δύναμη που θα παρτίζεται από 8.000 περίπου ε, στρατιώτες συν τους 5.000 στρατιώτες ε, του Μαλή, περίπου δηλαδή 13.000 ε, στρατιώτες που θα αναλάβουν την ασφάλεια της περιοχής. Άλλωστε τα στρατεύματα αυτά θα τα εκπαιδεύσουμε εμείς και όχι μόνο το στρατό του Μαλή, αλλά και άλλοι θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση των στρατιωτών από άλλες αφρικανικές ε, χώρες και οι Βρετανοί ε, ε, ασχολήθηκαν με την εκπαίδευση των στρατευμάτων του, της Νιγηρίας. Θα γίνουν παρόμοιες προσπάθειες, οπότε θα έχουμε μια στρατιωτική δύναμη αρκετά σημαντική που θα διαδραματίσει πολύ χρήσιμο ρόλο. Και άλλωστε μετά την Αφρικανική δύναμη αναμένεται και η δύναμη ε, διατήρησης της ειρήνης ε, των Ηνωμένων Εθνών. Και φυσικά χρειάζονται κάποιε εγγύσει για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού, αλλά και για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτών. Τώρα δεν ξέρω αν ε, θα αρκέσει αυτή η χρηματοδότηση, αλλά για, για να απαντήσω στη τελευταία ερώτηση της κυρίας Λέζινγκ, θεωρώ ότι αν θέλουμε μία γνήσια, μία πραγματική λύση για το μέλλον, όπως είπατε κι εσείς και αυτό επιθυμούμε, θα πρέπει να διερευνήσουμε και πολιτικές ε, λύσεις σε συμφωνία με την κοινότητα των Τουαρέγ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση. Οι αντάρτες, οι... Ε, μερικές δυνάμεις των ανταρτών μερικές φορές δεν είναι καν ε, ε, επίκοη του Μάιλι δεν είναι καν του ΑΡΕΚ. Μπορεί μερικοί να είναι το ΑΡΕΚ σε κάποιες ε, αντάρτικες ομάδες, αλλά στις ομάδες Ακμή και Ματζάου δεν υπάρχουν καν του ΑΡΕΚ. Ε, οι περισσότεροι αντάρτες προέρχονται από γειτονικέ χώρες. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των ανταρτών, που είναι κυρίως ένα φαινόμενο της μαφίας και της τρομοκρατίας και θα πρέπει να το εξαλείψουμε εκεί δεν επιδέχεται το θέμα καμία πολιτική λύση και έχουμε και την κοινότητα του ΑΡΕΚ που είναι κάτι τελείως διαφορετικό και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εκεί θα πρέπει να επιδιώξουμε μια πολιτική λύση. Τώρα αν αυτή θα λέγεται αυτονομία ή θα έχει άλλο όνομα θα αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Δεν θα επιβάλλουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαλί μια λύση για την εσωτερική κατάσταση. Και αν δούμε τι έκανε ο Νίγηρας πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, μετά κάποιες αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στις προηγούμενες συμφωνίες που είχαν συνάψει με την κοινότητα των Τουαρέκ, βλέπουμε ότι ε, διερεύνησαν και άλλες ε, λύσεις και τελικά φαίνεται ότι οι τελευταίες λύσεις είναι πολύ πιο επιτυχημένες από ό,τι προηγούμενες. Γιατί βάζοντα ΑΡΕΚ και στην κυβέρνηση και στο στρατό, γιατί ο πρωθυπουργό του Νίγηρα είναι το ΑΡΕΚ, ίσω εκεί θα ε, σημειωθεί πρόοδο τι θα είναι η διαφορά. Αλλά αυτό το αποφασίσουν ε, οι αρμόδιοι στο Μαλί. Δεν πρόκειται να, το να τους επιβάλλουμε εμείς ή να τους υπαγορεύσουμε μια λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκάλερ, θέλετε να συνοψίσετε. Όχι, μάλιστα. Περνάμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσίαση αυτή. Έχουμε τώρα δύο γρήγορα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο είναι η ενημέρωση από τους Κρίστιαν Νταν και τον Ντέβιν Μάρτιν σχετικά με την αποστολή παρατήρησης των εκλογών στην Ιορδανία. Κρίστιαν. Merci, merci infiniment. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Πρέντα και διακόπτη. Leave quietly the room so that... Παρακαλώ, παρακαλώ αποχωρήστε γρήγορα και ήσυχα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα αρχίσω, λέει ο κύριος Πρέντα, Έχω την εντύπωση ότι ο συνάδελφος David Μάρτιν δεν βρίσκεται εδώ, γιατί εκείνος ήταν ο βασικός παρατηρητής της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ήμουν επικεφαλής της μικρής ομάδας του Κοινοβουλίου που απαρτιζόταν από 7 μέλη. Κυρία Φαγιόν, Γκρίς, Μπουλάν, Βάικελ, Κόβαλε και Μπέλτερ. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τον συνάδελφο, τον David Μάρτιν και την ομάδα του. Να σας πω δύο λόγια για την αποστολή μας. Είχαμε εξαιρετικές επαφές κατά την διενέργεια των εκλογών με τις ε, ε, εκλογικές ε, αρχές της εκλογικής διαδικασίας και με τις δύο ε, Ισλαμικές ομάδες, κόμματα μάλλον, μέσα στα πλαίσια μιας διαδικασία αποκλεισμού που ίσχυε, ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και μετά είχαμε και τους μετριοπαθείς Ισλαμιστές που αποτέλεσαν και τη μεγάλη έκπληξη επίσης ένας υποψήφιος συνελήφθη μία μέρα πριν από την αφήξή μας διότι είχε εξαγοράσει ψήφους και ήρθαμε σε επαφή και με τον εκπρόσωπο της Συμμαχίας της Αριστεράς. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ καλή επιμελητιακή προετοιμασία ασχοληθήκαμε με τις εκλογές καθεαυτές στην Ιορδανία μέσα στα πλαίσια των ε, μεταρρυθμίσεων στη χώρα αυτή. Με τους, ήρθαμε σε επαφή με τους διάφορους φορείς. Είδαμε τις ε, πολιτικές ε, προοπτικές με περισσότερες επιφυλάξεις από πλευράς Ισλαμιστών Όσον αφορά την πλευρά των Ισλαμιστών, είδαμε και το θέμα της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Παλαιστινίων και εξελέγησαν 27 βουλευτές από τους 150. Υπήρξε ένα αναλογικό σύστημα, σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης, κάτι το οποίο οι Ισλαμιστές θεώρησαν ότι δεν ήταν επαρκές και ζήτησαν ακόμα πιο αναλογικό σύστημα. Τα ε, είδαμε και το περιφερειακά, ο, ε, περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα ως προς τη Συρία σχέσεις με τη Συρία και τις σχέσεις με το Ισραήλ. Οι εκλογές στο Ισραήλ διενεργήθησαν μία μέρα πριν από εκείνες της Ιορδανίας. Τέλος, ως προς την εκπροσώπηση των γυναικών, υπήρξε ένα 10% μια ποσόστοση 10% για τις γυναίκες και ίσως λίγο περισσότερο. Και μερικές επευλήθησαν πέρα από αυτή την ποσόστοση. Έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, αλλά αυτό αποτελεί ακόμα θέμα όπως και η ελευθεροτυπία. Πολλά θα πρέπει να βελτιωθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά την ευθύνη του τύπου για διάφορα σχόλια που ανακοινώθηκαν, που προωθήθηκαν. Επειδή είναι προχωρημένη ώρα και επειδή ο David Μάρτιν είναι εδώ πλέον και μπορεί να μας πει περισσότερα ο ίδιος, θα ήθελα να πω ότι κατά την ημέρα των εκλογών μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχε μια εκλογική εκστρατεία ακόμα και μπροστά στα εκλογικά κέντρα βεβαίως με ησυχία μεγαλύνει, χωρίς να έχει εκρηκτικό χαρακτήρα και είδαμε ότι υπήρξε πολύ καλή προετοιμασία του προσωπικού, καλή διοργάνωση, δεν είχαμε ατυχή συμβάντα. Και έτσι τα συμπεράσματά μας ήταν θετικά ως προς ε, αυτή την ε, ε, εμπειρία που είχαμε. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε αποστείλει παρατηρητές σε αυτή τη χώρα, στην Ιορδανία. Περισσότερο θα μας πει ο David Μάρτιν. Ο David Μάρτιν έχει το λόγο. chief observer of Ο επικεφαλής της Επιτροπή Παρακολούθησης. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Κρίστιαν. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία με το Κοινοβούλιο, με την ε, προσωπία του Κοινοβουλίου και την ε, Επιτροπή ε, παρακολούθηση ήταν εξαιρετική. Όπω ακούσατε, το πλαίσιο των εκλογών στην Ιορδανία μετά από κάποια χρόνια από την Αραβική Επανάσταση με, πόλεμο, με τον πόλεμο στα σύνορα με την Συρία και σε ό,τι αφορά τι ταραχές στο ιστορικό της χώρας για την ενέργεια και για τα τρόφιμα, για τις τιμές τους. Πολλά ήταν οι προσδοκίε ε, από τις εκλογές για την βελτίωση της δημοκρατίας και για την ε, υποστήριξη της Ιορδανίας για να εξέλθει από την κρίση. Οι εκλογές ήταν από τεχνικής άποψης πολύ καλά οργανωμένες. Οι ανεξάρτητοι εκλογική επιτροπή η οποία ιδρύθηκε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές λειτουργήσε εξαιρετικά και η ύπαρξή της επέτρεψε σε εμάς να παραστούμε με την αποστολή παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι, και πολύ το επισήμεναν, είναι ότι μπορεί να διοργανώθηκαν άριστα οι εκλογέ, αλλά τίποτα δεν άλλαξε στη χώρα μετά τις εκλογές, γιατί το εκλογικό σύστημα οργανώθηκε για να μπορέσουν ε, οι φυλέ να εκλέξουν ε, τα δικά του άτομα. Δεν υπήρξε άλλη αιτιολογία σε ό,τι αφορά την εκλογή των υποψηφίων. Ήταν ε, σχεδόν μοναδικό στον κόσμο Υπάρχει ένα σύστημα εκλογικό με μία ενιαία ψήφο μη μεταβιβαζόμενη σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα και 27 ήταν τα εθνικά κόμματα. Κανένα κόμμα δεν πήρε πάνω από δύο έδρες. Ήταν λοιπόν εξαιρετική η διοργάνωση των εκλογών. Εκλέχθηκαν 250 άτομα χωρίς όμως κάποια συγκεκριμένη εντολή, χωρίς κάποια συγκεκριμένη πολιτική που θα ακολουθήσουν. Η εκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από έλλειψη οικονομική κοινωνικού προγράμματος. Το θέμα ήταν μόνο να εκλεχθούν οι εκπρόσωποι της κάθε φυλής. Καλή αρχή λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, βελτίωση της δημοκρατίας στην Ιορδανία, γιατί να θυμόμαστε το 2010 οι μυστικές υπηρεσίες ε, στην Ιορδανία ε, παραδέχτηκαν ότι είχε γίνει νοθεία στις εκλογές. Τώρα αυτή τη φορά δεν το παραδέχτηκαν ότι το είχαν πράξει οι ίδιοι, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι δεν συνέβη. Σε επόμενη φάση θα πρέπει να κοιτάξουμε τα πολιτικά κόμματα, την χρηματοδότησή τους, προκειμένου να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, προκειμένου να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αναγνωρίσει ο κόσμος και θα το υπερψηφίσει. Άρα, Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή αρχή από πλευρά τη διοργάνωση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θέλει κανεί το λόγο, Όχι. Κύριε Πρόεδρε, μερικές παρατηρήσεις ε, που σε παρατηρήσει εκλογών σε χώρες σαν την Ιορδανία ε, είναι κάπως ε, εντυπωσιακές όπως είπε ο κύριος Πρέντα, η προεκλογική εκστρατεία κράτησε μέχρι και την ημέρα των εκλογών μπροστά στις κάλπες. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε όμως. Είναι ε, αρκετά συγκλονιστικές αυτές οι παρατηρήσεις γιατί δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κουλτούρα. Υπήρχαν παρατηρητές και από τα πολιτικά κόμματα αλλά και από οργανώσεις που ασχολούνται με την παρακολούθηση τη της δημοκρατικής διαδικασίας εντός της Ιορδανίας. Και αυτό ήταν ενδιαφέρον λοιπόν. Επίσης ε, εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ε, στην η Επιτροπή ε, στα εκλογικά τμήματα είχαμε ξεχωριστά εκλογικά τμήματα για γυναίκες και ξεχωριστά για άντρες. Ενώ στην, ε, στις εκλογικές επιτροπές ήταν ανάμεικτη η σύνθεση και ανδρών και γυναικών. Υπήρχαν και σε εκλογικά τμήματα που για γυναίκες ε, μέλη της Επιτροπής της ε, Φορευτικής που ήταν και άντρες. Και αυτό ήταν κάπως περίεργο. Επίσης, ε, οι εκλογές σε τέτοιου είδους χώρες ε, έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Σε κάποια εκλογικά τμήματα, ε, σε εκλογές με πλειοψηφικό σύστημα, είχαμε γυναίκα υποψήφιο, σε εκλογικό τμήμα που μόνο γυναίκες και εκεί μόνο τρεις ψήφους έλαβε. Θέσαμε λοιπόν ερωτήσεις και απορίες στους συνομιλητές μας από την Ιορδανία. Πώς σχολιάζουν τέτοιου είδους εκλογές. Φανταστήκαμε ότι θα ίσχυε μια γυναική αλληλεγγύη σε εκλογικό τμήμα με αποκλειστική συμμετοχή γυναικών, να ε, υπάρχει υποψήφια γυναίκα και να μην την ψηφίζουν οι γυναίκες. Αλλά μας είπαν ότι περισσότερο αποφασιστική σημασία έχει στην Ιορδανία ε, το θέμα του οικογενειακό παρά το θέμα του φίλου. <laughs> Ενώ στην ε, ευρωπαϊκή κουλτούρα έχουμε και άλλου είδους αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Κάτι άλλο ενδιαφέρον που παρατήρησα ήταν ότι στην παρατήρηση εκλογών ε, σε παραδοσιακές τοποθεσίες όπου μένουν κάποιοι γηγενείς Ορδανοί ή σε άλλες περιοχές που κατοικούνται από πολυπληθείς ομάδες Παλαιστινίων που μπορεί να γεννήθηκαν στην Ιορδανία αλλά το, η ιδιοσυγκρασία τους είναι πολύ διαφορετική και η συμπεριφορά τους είναι πολύ διαφορετική. η εξωτερική, η εξωτερήκευση αυτή τη συμπεριφορά στην εκλογική μέρα είναι διαφορετική μεταξύ Παλαιστινίων, για παράδειγμα, και Γηγενών ε, Ιορδανών. Όπω είπε και ο κύριο Πρέντα, η εκλογική διαδικασία λαμβάνει πολύ καλή βαθμολογία, είναι πολύ θετική η αξιολόγηση. Έχουμε ενιαίο σύστημα καταγραφής των, των ψηφοφόρων και μάλιστα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να διδαχθούν ε, από αυτό το σύστημα και μάλιστα είχαμε και οπτικό, οπτική απεικόνηση του ψηφοφόρου, όπου, ώστε η Εφορευτική Επιτροπή μπορούσε να ε, εξακριβώσει κατά πόσο ο ψηφοφόρος που είχε προσέλθει στην κάλπη είναι αυτός που αφαινόταν στην, ε, στην οθόνη και στις φωτογραφίες. Εντυπωσιακό λοιπόν αυτό το σύστημα καταγραφής. Υπήρξαν βέβαια και κάποιες μικρές ε, ατασταλίες, αλλά επαναλαμβάνω το θέμα της, κεντρικής, της ενιαίας καταγραφής με την Κεντρική ε, Εκλογική Επιτροπή ήταν πολύ εντυπωσιακό και σωστό. Σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας. Είναι νομίζω σημαντική η ενημέρωση αυτή. Θα μας υποβάλλετε και σχετικό έγγραφο για την προετοιμασία της Ορδανίας σε ό,τι αφορά και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέσουμε και τα βασικά ερωτήματα που θα ανακύψουν από τα απορίσματα που θα μας υποβάλλεται. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση αυτή, κοιτώντα και την κατάσταση στις αραβικές χώρες και στην Αφρική. ο, ο δρόμος της Επανάστασης είναι ο σωστός δρόμος και κοιτώντα την Ιορδανία βλέπουμε ότι ο δρόμος του εκδημοκρατισμού χαρακτηρίζεται και από πολλές διαφορές και σε ό,τι αφορά το σημείο κίνησης, τον, τη μεθοδολογία που ακολουθείτε, αλλά και το αποτέλεσμα που προκύπτει. Θεωρώ ότι η Ιορδανία μας δίνει ένα σημαντικό, μια σημαντική απάντηση. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης της σημερινής. Η κυρία Γκόμες μας ζήτησε να το αναφέρουμε εν συντομία. Δεν έχουμε χρόνο για λεπτομέρειες να δώσουμε στην συνάδελφο να αναφέρει το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά την ανάκτηση δεσμευθέντων περιουσιακών στοιχείων δικτατόρων κτλ. Στην ε, Αραβική Επανάσταση. Η Άννα έχει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι στη συνάντηση που είχαμε στην Κύπρο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο Μπερνάρντιν Ελιόν ε, ρώτησε τους ευρωβουλευτές ε, κατά πόσο θα μπορούσαν να μειχθούν και μας ζήτησε μάλιστα να, να πρωτοστατήσουμε σε κάποιες πολιτικές δράσεις και να συνεργαστούμε με τις χώρες Αραβικής Άνοιξης για την ανάκτηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Και είπε ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα γίνουμε περιζήτητος εταίρος και για τις κυβερνήσεις των χωρών της Αραβικής Άνοιξης αλλά και για τους λαούς των χωρών αυτών. Έτσι, η ομάδα μου οργάνωσε ένα σεμινάριο ανοιχτό προς όλους, στείλαμε προσκλήσεις ε, προς όλους και χαρήκαμε ιδιαίτερως γιατί οι πρεσβείες της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τινησίας έλαβαν μέρος στο σεμινάριο αυτό και στην περίπτωση μάλιστα της Τινησίας είχαμε και εμπειρογνώμονες ε, υψηλού επίπεδου από την ε, Ειδική Επιτροπή που συστήθηκε την Ισία για την ανάκτηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Στο σεμινάριο συμμετείχε και η Ελβετία, γιατί η Ελβετία είναι από τις χώρες ε, στις οποίες έχουν μπλοκαριστεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Και ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τη δικτατορία του Μάρκος στις Φιλιππίνες ε, για να ανταποκριθεί στις αιτήσει ανάκτησης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Οπότε υπήρξε κάποια δράση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν θέλετε να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πίνο Αρλάκη που διατύπωσε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό και είπε ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από την ΕΙΕΔ να συστήσει ε, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συνδράμει με νομική εμπειρογνωμοσύνη στα περίπλοκα ζητήματα που ανακύπτουν και που δεν είναι μόνο πολιτικά αλλά είναι κυρίως νομικά. Γιατί θα πρέπει να συνοηθούμε με τους εμπειρογνώμονες των χωρών της Αραβικής Άνοιξης για να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα νομικά, οι νομικές πτυχές. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο αυτό το σημείο, γι' αυτό και ζήτησα να συμπεριληφθεί στην ημερήσια μας διάταξη. Εμείς πάντως σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις γνώσεις που έχουμε θα μπορούσαμε και έθεσα το αίτημα στη διάσκεψη των Προέδρων και ίσως ε, στην επόμενη Ολομέλεια ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα έχουμε και συζήτηση με ψήφισμα ζητώντας από την ΕΙΕΔ να μας ενημερώσει τι έκανε και πώς ε, έλαβε υπόψη τις προτάσεις ε, του Πίνο Αρλάκη. Κυρία Νέιτς, πρόεδρε, να επανέλθουμε στο θέμα αυτό αν θα θέλατε στην επόμενη συνεδρίαση όταν θα είναι και πιο πολλοί βουλευτές εδώ στην Επιτροπή γιατί δεν νομίζω ότι είναι ότι είμαστε αρκετοί για να λάβουμε την οποιαδήποτε απόφαση για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Άκουσα με προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε σύσταση στην παρούσα φάση. Επειδή δεν είναι αρκετοί συνάδελφοι που είναι εδώ. Να το συμπεριλάβουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Όχι πως ε, δεν ε, είμαστε λίγοι και καλοί, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η ποιότητα δεν μπορεί να καλύψει την έλλειψη ποσότητας. Ναι, αυτό είπα και εγώ εισαγωγικά λέει ο Πρόεδρος. Αυτό είπα στην Άννα, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, σημειώνεται ε, ένα λάθος στην ημερήσια διάταξη. Επόμενη συνάντηση της Επιτροπής είναι την 5η στις 9 μαζί με την ΣΕΝΤΕ. Να σας το υπενθυμίσω αυτό γιατί αναφέρεται ότι η επόμενη συνεδρία είναι τη Δευτέρα. Είναι παλαιότερη, παλαιότερο σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Thank you. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι αύριο το απόγευμα είμαστε όλοι προσκεκλημένοι στη δεξίωση της Λέτης Άστον. She Μας υποσχέθηκε πολύ καλό κόκκινο αγγλικό κρασί.